για τη μείωση των εκπομπών και τι μπορούμε να κάνουμε στην χρηματοδότηση άλλων χωρών. Μακροπρόθεσμα, πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ενδεχόμενο μόνιμης χρηματοδότησης κάποιων μέτρων, αλλά στην προκείμενη στιγμή η άμεση χρηματοδότηση είναι αυτή που επήγει. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τους μηχανισμούς αγοράς μας για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε κεφάλαια και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, όσων έχουμε ήδη πράξει. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι έγινε, για παράδειγμα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τις τεχνολογικές τροποποιήσεις. Τον Ιούλιο είχαμε μια άτυπη σύνοδο υπουργών που μας επέτρεπε να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει να τονίσω ότι έχουμε σημαντική υποστήριξη, πολιτική υποστήριξη από κάθε πλευρά στο τομέα αυτό. Επίσης θέλουμε η μείωση 20 με 30% να, από 20 30% να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός περαιτέρω αλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διαθέτουμε ένα στέρεο ε, τεχνικό εργαλείο. Έχουμε προχωρήσει μια σειρά πρωτοβουλειών για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τους εταίρους μας και έτσι, πριν το καλοκαίρι ξεκινήσαμε διαπραγματεύσει με την Κίνα και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην επόμενη σύνοδο Κορυφή θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα ε, εν ώψη της Κοπενχάγης που αποτελεί ένα κλειδί, ένα σημείο κλειδί για τις περαιτέρω εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τις εθνικές κυβερνήσεις και με τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πλονεκτήματα των αλλαγών. Μία οικολογικά αποδοτική οικονομία τώρα, το δεύτερο τομέα. Στον τομέα αυτό η Προεδρία έχει επίγνωση τη υφιστάμενη οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η κρίση αυτή θα πρέπει να μα πρόξει ακόμα περισσότερο προ την κατεύθυνση οικολογική κουλτούρα. Αυτή η οικολογικά αποδοτική οικονομία απετέλεσε αντικείμενο των συζητήσεων που είχαμε κάνει σε μια κοινή σύνοδο Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Εδώ είχαμε τονίσει ιδίω την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευθύνες συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να κινητοποιήσουμε τον πληθυσμό. Στο επίπεδο αυτό υπογραμμίσαμε ιδιαίτερα τις οικονομικές πτυχές του θέματος. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε τις ε, βλαβερές προς το, επιβλαβείς προς το περιβάλλον ενισχύσεις. Το φθινόπωρο θα ασχοληθούμε λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία της Λισαβόνας, προσπαθώντας να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε την οικονομία μας, ούτως ώστε να μετατραπεί σε μια οικολογικά αποδοτική ευρωπαϊκή οικονομία. Και ξέρουμε, έχουμε πραγματική επίγνωση ότι μπορούμε να στηριχτούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βιοπικιλότητα. Στο θέμα αυτό χρειάζεται να θέσουμε νέους διεθνείς στόχους που θα είναι περισσότερο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την προστασία της βιοπικιλότητας. Στη Σουηδία οργανώσαμε ήδη κάποιες ε, ε, συναντήσεις σχετικά, προσπαθώντας να υιοθετήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για να καλύψουμε τις φιλοδοξίες μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εν ώψη του 2000, πέραν από το 2010. Ε, δίδουμε μεγάλη, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο τι μπορούμε να κάνουμε ε, για την κοινωνία, γιατί η κοινωνία θα το πληρώσει αν καταστραφούν κάποιοι βιότοποι, κάποιες, ε, κάποια είδη πανίδας ή χλωρίδας. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία που θα βελτιώσει την κατάσταση στην κοινωνία μας. Το κείμενο αυτό, το Visions for Diversity Beyond 2010, είναι ένα κείμενο το οποίο νομίζω θα βοηθήσει να προχωρήσουμε. Όταν μιλάμε για την βιοπικιλότητα, θα ήθελα να σας πω ότι η χώρα μου ε, είναι ικανοποιημένη από τις προτάσεις που έγιναν για να για να υιοθετηθεί μια διεθνής πλατφόρμα ανταλλαγής ε, ε, βέλτιστων πρακτικών που ελπίζουμε να τεθεί σε λειτουργία του χρόνου. Και περιμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα του τι μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε με καλύτερο τρόπο την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ενάλλειο πλούτο, η θάλασσα είναι πολύ σημαντική για την οικονομία μας. Ξέρουμε ότι κάθε περιοχή είναι μοναδική και στο επίπεδο αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι, έχουμε κάνει σε κάθε τομέα για να μπορέσουμε φερρυπίν να έχουμε μία πιο υπεύθυνη αλίευση κάποιων ειδών. Η πολιτική για τη θάλασσα είναι σημαντική για τον καθένα μας. Επιπλέον υπάρχουν και ορισμένε φιλοδοξίες σε περιφερειακό, κάποιοι στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικοί για την επίτευξη των συνολικών στόχων. Το Δεκέμβριο θα έχουμε μια πολύ σημαντική ε, συνάντηση για το θέμα αυτό. Ε, Ιδίω ό,τι αφορά την στρατηγική για την ε, περιοχή της Βαλτικής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν κάποιες περιφερειακές ή κάποιες παγκόσμιες προσεγγίσεις για να λύσουμε παγκόσμια ή περιφερειακά προβλήματα αντίστοιχα. Πρέπει ταυτόχρονα να μπορούμε να λάβουμε υπόψη και άλλες διαστάσεις. Την ε, γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλληλεία. Πρέπει να έχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση. Η Επιτροπή στο σημείο αυτό έκανε μια σειρά προτάσεων οι οποίες προσπαθούν να εξετάσουν τι συνέπειες θα έχει φερκίνη απαγόρευση αλίευσης κάποιων ειδών. Αν η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι. Όπως σας είπα η περιοχή της Βαλτικής που είναι ένα παράδειγμα για μας είναι μια πολύ ευαίσθητη ε, βιολογικά περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τομέα αυτό είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει. Υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα intergroup για την Βαλτική που μπορεί σίγουρα να παίξει έναν κεφαλαιόδου σημασία ρόλο στην συζήτηση του μέλλοντος της θάλασσας αυτής. Θέλουμε, πιστεύουμε μάλλον ότι η δουλειά στον τομέα της Βαλτικής θα αποτελέσει έμπνευση για την Επιτροπή ούτως ώστε να αντιμετωπίσει με παρόμοιο ή με, με ομοιόμορφο τρόπο και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε νομοθετικό επίπεδο τώρα, τον τελευταίο καιρό, είχαμε μια σειρά νέων προτάσεων σε επίπεδο περιβάλλοντος προσπαθήσαμε να εξετάσουμε ποιος θα ήταν ο ρόλος της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να στηριχθούμε στη βοήθεια του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα δηλαδή της Επιτροπής σας και ελπίζουμε να μπορέσουμε μαζί να προετοιμαστούμε για τις μεγάλες διεθνείς συναντήσεις που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει και η οδηγία για τα απόβλητα, βέβαια ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό κείμενο, καθώς και η οδηγία για τους περιορισμούς της χρήσης κάποιων επικίνδυνων προϊόντων η, οδηγία για τα βιοκτώνα προϊόντα και ελπίζουμε να επανέλθουμε προχωρώντας και σε άλλα νομοθετικά κείμενα όπως η οδηγία για τα βιομηχανικά απόβλητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι περιμένω με ανυπομονησία τις ε, απόψεις και τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να τις θέσετε. Παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Herr uh, uh, Andreas uh, Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση του προγράμματος ε, της ε, Προεδρίας σας σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοπικιλότητα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ε, και όλες τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες επίκυνται στο εγγύης μέλλον. Υπάρχουν βέβαια συνάδελφοι τώρα που έχουν ζητήσει το λόγο. Και να πω βέβαια πριν δώσω το λόγο εδώ στους άλλους ομιλητές πώ και η Επιτροπή μας αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία με τη δική σα Προεδρία και είμαστε σίγουροι πω θα έχουμε ε, θετικά αποτελέσματα. Ο κύριο Ζέμα, έχει το λόγο. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σα, παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σα ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή με την πρόθεση να συζητήσετε ε, αυτά τα ζητήματα μαζί, μαζί μα και βέβαια εμεί θα υποστηρίξουμε από πλευρά τη δική μα Επιτροπή πλήρω τι δικέ σα προσπάθειε σε ό,τι αφορά το πακέτο για το κλίμα και την διάσκεψη στη Κοπενχάγη. Ε, αποφασιστική σημασία για την ε, επιτυχή έκβαση αυτή τη διάσκεψη θα είναι φυσικά ο καθορισμό δεσμευτικών στόχων. Ε, όχι όμω μόνο αυτό ο καθορισμό των δεσμευτικών στόχων, αλλά και η θέσπιση ενός μηχανισμού επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τους στόχους που έχουν θέσει στους εαυτούς τους. Ε, νομίζω πως αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης, δηλαδή ε, ποιες δυνατότητες θα έχει η διεθνή κοινότητα να κινηθεί κατά κρατών, μελών, τα οποία, ε, κρατών συγγνώμη, τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρήσουν ορισμένους στόχους, αλλά δεν ε, τελικά δεν το έχουν πράξει. Γιατί έχουμε δει από την εμπειρία μα ότι ε, υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το επίπεδο και βέβαια ε, κυρίως αναφέρομαι εδώ στι χώρε πριν. Δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, ε, Κίνα και ούτω καθεξής οι οποίε ε, ε, από τη μία πλευρά θέλουν να τη χάνουν μεταχείριση στι αναπτυσσόμενε χώρε, από την άλλη ισχυρίζονται ότι δεν είναι πλέον αναπτυσσόμενε χώρε. Οπότε ε, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια ομάδα κρατών τα οποία έχει το δικό τη σημαντικό μερίδιο σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και η οποία δεν θέλει τόσο να ε, συμμετάσχει στον καθορισμό τέτοιων ε, δεσμευτικών ε, στόχων σε ό,τι αφορά την μείωση τη ρήπανση και ταυτόχρονα ενδεχομένω δεν θα θελήσει να προβεί και στην υπογραφή μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει και μηχανισμό επιβολή κυρώσεων για τη μη στόχων. Τι θέλετε λοιπόν να κάνετε από την πλευρά τη δική σα Προεδρία. Από εκεί και μετά έχουμε να κάνουμε βέβαια και με την με τα την ε, μετάθεση, αν θέλετε, ε, πόρων. Αλλά εδώ δεν αναφέρομαι μόνο σε χρηματικού ε, πόρου. Εκείνο που μα ενδιαφέρει είναι η μεταβίβαση τεχνολογικών πόρων, τεχνολογία. Δηλαδή, οι μέχρι τώρα εξελίξει στον χώρο τη πολιτική έχουν καταδείξει, κατά τη δική μα γνώμη, ότι πολλέ φορέ η απλή μεταβίβαση οικονομικών, χρηματοδοτικών πόρων τελικά δεν καταλήγει εκεί που πρέπει. Δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει αυτοί οι πόροι. Οπότε, με ποιο τρόπο θέλει η Σουδική Προεδρία να οργανώσει τη μεταβίβαση τεχνολογικών πόρων χώρων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη που ε, λαμβάνουν αυτούς τους πόρους να μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ώστε να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών. Ένα ακόμα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον. Να πω λοιπόν πως οι σημαντικότερες επιπτώσεις ε, των κλιματικών μεταβολών ε, πρέπει να αναμένονται στο μέτωπο, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, εντό εισαγωγικών, της θάλασσας. Οπότε ε, θα πρέπει να αναλάβουμε ε, και εδώ μια αυξημένη ευθύνη δηλαδή του να έχουμε μια ε, ευρύτερη παγκόσμια θαλάσσια πολιτική σε ό,τι αφορά τις κλιματικές μεταβολές. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, τον κύριο Ζέμπα. συνάδελφος. Um, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε. Θα είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσει για τους στόχους της ε, πολιτικής για την προστασία του κλίματος. Ξέρουμε ότι τα ΙΠΑ έχουν προτείνει κάποιους στόχους. Στη σχέση το 2005 φαίνονται φιλόδοξοι αυτοί οι στόχοι. Όμως σε σχέση με τους δικούς μας στόχους, μάλλον ε, συγκρατημένοι είναι αυτοί οι στόχοι, μάλλον ε, μέτρη είναι. Άρα για πες μας πώς τα βλέπετε εσείς δεύτερον. Για σχέση με αυτό που έγινε στην Αυστραλία και στο κοινοβούλιο εκεί πέρα. Γιατί το σύστημα εμπορίας των εκπομπών. για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό ήταν όλη η κουβέντα. Πώς θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο είδους ε, πρότυπα, κάποιο είδους κανόνες που θα πρέπει να θεσπιστούν ούτως ώστε να μην έχουμε ε, διπλές καταμετρήσεις. για την αντιστάθμιση που θα γίνεται δηλαδή σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι τον έχουμε κάποιον σχετικό μηχανισμό. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο σχετικά με αυτό. Κρίς. Κρίς Ντέβις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω κύριε Υπουργέ για την Κοπενχάγη πρώτα. Κάτι θα βγει από τις διαπραγματεύσεις. Θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία γιατί φαντάζομαι θα είναι ντροπή να φύγουμε από εκεί χωρίς να έχουμε τίποτα στις βαλίτσες. Το θέμα είναι κατά πόσο βέβαια αυτό που θα συμφωνηθεί θα έχει κάποια αξία, απλώ θα είναι και ένα λόγιο. Δεύτερη ερώτηση. Έχω δέκα χρόνια σε την επιτροπή, ξέρω ότι θεσπίζουμε ένα σωρό νομοθετήματα, αλλά πολλέ φορέ το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται αυτά τα οποία θεσπίζουμε. Όλοι έχουν παραδείγματα τέτοια σε όλε μα τι χώρε. Πάντοτε απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτάμε γιατί δεν εφαρμόζονται τα μέτρα, λέμε για ποιο λόγο η διαδικασία πάντοτε τη εκτέλεση τόσο βραδία. Γιατί δεν με μια πιο πολιτική διαδικασία αντί να περνάμε μέσα από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Για πέστε μας στο Συμβούλιο πόσο συχνά σας απασχολεί το θέμα της ε, εφαρμογής των νομοθετημάτων. Για... Ε, θα υπάρχει σήμερα στη διάταξη αυτό το θέμα για αυτή την Προεδρία ή για την επόμενη. Ή ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Ε, εσείς την Κομισιόν και η Κομισιόν εσάς. Ότι δεν κάνει ο καθένας καλά τη δουλειά του. Έχει φυσικά πάρα πολύ καλές επιδόσεις στη Σουηδία στα σχετικά θέματα. Επομένως, δικαιούται να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. ούτω ώστε να μην χρησιμοποιούνται νομικά μέσα, αλλά μάλλον πολιτικά για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θα κάνετε τέτοιες κινήσεις κατά αυτή ε, την Προεδρία σας. Σαν του Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. μπορούσε να είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να καταλάβουν οι χώρες αυτές ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα να τα πούμε. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Αναφέρεται στην ε, στο σελίδο 2, ως προτεραιότητα η Προεδρία σας θέλει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον Ιδράργυρο. Πέστε μας δύο λόγια παραπάνω. Με ποια διαδικασία θα προχωρήσετε. Νομοθετικές προτάσεις θα κατεβάσετε. Πώς θα σημειώσετε κάποια πρόοδο σε αυτό το θέμα, σε αυτό το μέτωπο. Επίσης υπάρχει κάποια ε, πρόταση για τις εκπομπές διοξιδίου όσον αφορά τα, τα βάντα, τα, τα μικρά φορτηγάκια, τα μίνι λεωφορεία. Υπάρχει επισυνόηση με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για θέσπιση κάποιας νομοθεσίας. And de Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό. Βιοπικιλότητα. Θέλω να ρωτήσω. Σωστά αυτά που είπε ο κύριος Υπουργό για την συνάντηση στο Στρόμσεντ και την πρόταση για την Διεθνή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Βελτιστών Πρακτικών. Ωστόσο, τι θα κάνετε κύριε Υπουργέ με σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες προτάσεις. Τι προτάσεις θα υποβάλλετε δεδομένου της έλλειψης, της μη υλοποίησης του προγράμματος δράσης για τη βιοπικιλότητα και των έντονων πιέσεων που δεχόμαστε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων, όχι μόνο την ε, διακοπή της μείωσης της βιοπικιλότητας. Προτείνω να κάνετε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων κύριε Υπουργέ αν θέλετε και μετά να ξαναγυρίσουμε. So, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με τα ερωτήματα που λέω του κ. Ρίτσαρτ Σίμπερ. Σε ό,τι αφορά Ε, αυτό που είπατε ε, σε σχέση με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, τις αναδυόμενες οικονομίες. Ναι, θα πρέπει να έχουμε υψηλές αξιώσεις από αυτές και το είπαμε με πολύ σαφή τρόπο, για παράδειγμα, προς την Κίνα, Κάτι τη συνάντηση Τρόικα στο Πεκίνο. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες αξιώσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών BRIC. Και φυσικά ταυτόχρονα συζητήσαμε τη φύση ε, αυτή τη προβληματική του να δημιουργηθούν δηλαδή δεσμεύσει, δεσμευτικοί στόχοι, γιατί προφανώ και είναι σημαντικό. Ε, και ε, όπως το εκφράσαμε αυτό στην Κίνα, μας είπε ότι υπάρχει μια ισχυρή εθνική νομοθεσία, αλλά αυτό που θέλουμε εμεί να κάνουμε είναι να διασυνδεθεί αυτή η εθνική νομοθεσία με μια διεθνή συμφωνία. Προφανώ βρισκόμαστε ακόμα σε φάση συζήτηση με την Κίνα και με άλλου. Ε, και με τις ΗΠΑ και με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ως προς το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια τέτοια σύνδεση. Αλλά ε, ε, αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή του να υπάρξει μια διασύνδεση των εθνικών δεσμευτικών στόχων ίδια ε, διατάξεων με ε, ένα διεθνές πλαίσιο, μια διεθνή συμφωνία που θα ε, ακριβώς μεταφέρει αυτούς τους στόχους, αυτές τις εθνικές δεσμεύσεις στο διεθνές επίπεδο. Να μην υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, θα προωθήσουμε αυτό το ζήτημα, θα αποτελέσει δηλαδή το, το στοιχείο της δέσμευσης ένα βασικό στοιχείο σε μια ε, μεταγενέστερη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, παρακολούθηση και τις χρηματοδοτικές ε, ροές και την εποπτεία τους, είναι πράγματι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο του πώς θα δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη ΣΥΕΜ ως ένα παράδειγμα. Θα εδώ έχουμε λοιπόν ένα σύστημα από την πλευρά των ΗΠΑ για τον έλεγχο. Ε, και, ε, να, και απαντώντας εδώ και στην Λίνα Μακέμπαν, δηλαδή πραγματικά είναι σημαντικό εδώ να έχουμε υψηλότερα πρότυπα για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, τα, ε, την ε, κατάλληλη ποιότητα και στο πλαίσιο συμφωνιών όπως αυτή η CEM. Και εμείς από την πλευρά μας προωθούμε ένα τέτοιο μηχανισμό και μέσα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος CEM στο οποίο συμμετέχουμε. Κάτι τέτοιο όμως ισχύει γενικότερα και για το ζήτημα των, της μεταφοράς τεχνολογικών πόρων, δηλαδή τεχνολογίας και ούτω καθεξής. το σημείο της αφετηρίας είναι η ε, μακροπεριφερειακές ε, πολιτικές. Άρα λοιπόν αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να προωθήσουμε την ε, δική μας πολιτική για την Βαλτική κατά τη δική μας προεδρία, ούτως ώστε να αποτελέσει το παράδειγμα για τη δουλειά για άλλου τέτοιου είδους μακρο project και στην ε, διάσκεψη του Δεκεμβρίου θα έχουμε ε, τέτοια παραδείγματα από το χώρο της Μεσογείου, από, τον, ε, από τις χώρες του Δούναβε, από τον χώρο της Μαύρης Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και τέτοιου είδους παραδείγματα θα μπορούσαν να συνδεθούν και στο ευρύτερο επίπεδο, ε, με το ευρύτερο επίπεδο της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής της Ένωσης δηλαδή, αλλά και με το διεθνές επίπεδο. Λέντε, τώρα σε σχέση με αυτό που είπες ως ε, προς τα όσα αναμένουμε από τους Αμερικάνους. Εγώ είχα την δυνατότητα σε διμερές επίπεδο να εκφράσω τις δικές μας προσδοκίες έναντι τους και μάλιστα ε, με μια τέτοια συχνότητα που μερικές φορές είχα την αίσθηση ότι είχαν αρχίσει να κουράζονται με, την, ε, με τις δηλώσεις μου σε σχέση με τα όσα δηλαδή αναμένουμε εμείς από την πλευρά τους. Εκείνο που θα είναι αποφασιστικό είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε να δείξουν ότι μπορούν να βρουν ένα μονοπάτι, μια οδό προ τη μείωση των εκπομπών που πράγματι να μα πείσει αξιόπιστα ότι θα ε, επιτύχουν ε, το στόχο ε, τη μείωση των δύο βαθμών. Θερμοκρασία δηλαδή. Ε, Μα είπαν πω υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά θα θέλαμε να δούμε πώ θα το επιτύχουν. Δηλαδή να επιτύχουν τον αντίστοιχο στόχο για τη δική του χώρα, σε εθνικό επίπεδο, για να δούμε τελικά για να μπορούμε να δούμε και να καταφέρουμε από την πλευρά των αναπτυγμένων χωρών τα όσα θα πρέπει να επιτύχουμε σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών. Ε, και σε σχέση με το τελευταίο σημαντικό ε, σημείο που θέσατε σε ό,τι αφορά την Αυστραλία, ναι, πράγματι αποτελεί ένα βήμα ε, προς τα πίσω. Αναμένω τώρα από το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας να προβεί σε νέα βήματα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση εθνικής νομοθεσίας πριν από την διάσκεψη της Κοπεχάγης και ε, ε, το ανέφερα αυτό ε, στον συνάδελφό μου, στον ομόλογό μου από την Αυστραλία. Και είχαμε ήδη συναντήσεις και στην Ουάσιν και θα το κάνουμε στο μέλλον. Τώρα, Χριστέβη, σε ό,τι αφορά το σημαντικό ερώτημά σας το τι θα πρέπει να αναμένουμε από τη διάσκεψη της Κοπεχάγη. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής εδώ. Ε, καταρχήν, εκείνο που θα πρέπει να αναμένουμε είναι μία συμφωνία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ή να πληρεί ή να δώσει μία πλήρη απάντηση στους δύο στόχους που έχουμε. Ε, κατά δεύτερον, εκείνο που είναι επίσης σημαντικό είναι όλες οι χώρες να συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη, σε αυτή τη δέσμευση. Και ε, επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης γιατί αυτό που είδαμε ε, μέχρι στιγμής είναι ότι ε, κάθε, με κάθε νέο βήμα που έκανε η επιστήμη αυξήθηκαν και οι αξιώσεις, αυξήθηκαν δηλαδή και τα όσα αναμένουμε, όλες οι προσδοκίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιτρέπει και μια τέτοια δυναμική, μια συμφωνία που υιοθετηθεί για να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης ούτως ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι δικές μας ενέργειες πάντα συνάδουν με τα όσα επιβάλλονται από την επιστήμη. Σε ό,τι αφορά τα τώρα και την ε, σύστημα εμπορίας εκπομπών και ούτω καθεξής, προφανώς ε, και αναμένουμε με ενδιαφέρον εδώ και την ε, συζήτηση που θα γίνει και στο υπουργικό επίπεδο με τους ομολόγους μου. Η Επιτροπή, λόγω των συνδικών έχει ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση και την ε, επιβολή της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ποιες είναι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τι μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, αναγνωρίζουμε αυτήν την ε, νομική της αρμοδιότητα, από την άλλη πλευρά θα θέλαμε να έχει και αυξημένη αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις και, να, και του να παρέχει σε εμάς τους πολιτικούς ε, πληροφορίες στοιχεία προς το πώς ε, έχουν ποιο ήταν ο αντίκτυπο των πολιτικών. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει τόσο εργαλείο άσκηση πολιτική πίεση, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω συζήτηση τη πολιτική. Οπότε κάτι τέτοιο θα το αξίωνα. θα το χάσει. Ε, θα ήθελα πολύ να σας απαντήσω ε, ε, στα σουηδικά. Αλλά επειδή είχα αποσχεθεί ότι θα απαντώ στα αγγλικά, αυτό θα κάνω. Θα απαντήσω στα αγγλικά. ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Η Προεδρία, ναι, έχει την πρόθεση να το πράξει αυτό. Και Έχω μέχρι στιγμής λάβει την εντολή από τους ε, συνάδελφους ε, στο υπουργικό επίπεδο. Ε, ποιο θα είναι το πρώτο βήμα να επιδείξουμε ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Upfront financing. Και τώρα προσπαθούμε εδώ να έρθουμε σε επαφή με άλλους εμπλεκόμενους, με άλλους φορείς οι οποίοι και εκείνοι να ενεργοποιηθούν περισσότερο σε ό,τι αφορά τη χρωματοδότηση ούτως ώστε να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια έως το 2012-2013 που θα υπάρξει νέα πλέον συμφωνία και για να ε, διασφαλιστούν οι πόροι για τη δημιουργία περαιτέρω δυνατοτήτων ε, ε, δυνατοτήτων, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά των ε, συγκεκριμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μιας αρχιτεκτονικής, μιας δομής που θα καλύπτει όλο το χώρο της χρηματοδότησης. Εγώ αναμένω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έχει μια πλήρη εικόνα του πώς θα δημιουργηθεί μια τέτοια δομή πριν από την ε, διάσκεψη της ε, Κοπενχάγης. Και εδώ συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι και εκείνοι θα είναι έτοιμοι για τη συζήτηση της διάσκεψης. Και επιτρέψτε μου να πω πως καθώς προετοιμάζουμε το μηχανισμό της χρηματοδότησης θα πρέπει να διερωτηθούμε ευθύ εξ αρχής από πού απορροφώνται αυτοί οι πόροι. Πού κατευθύνονται. Και υπάρχουν ε, δημόσια κονδύλια τα οποία θα χρειαστούν και τα οποία ε, θα κατευθυνούν και πέρα από την άμεση απευθεία ε, βοήθεια και σε άλλους τομείς και ταυτόχρονα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε και ιδιωτική συγχρηματοδότηση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και άλλα ενδιαφέροντα ε, projects. Και γι' αυτό ε, λέμε με τόσο εμφαντικό τρόπο ότι αναμένουμε να λάβουμε επιτάπητο στις προτάσεις από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών τους ώστε να ε, διασφαλίσουμε ότι το σύστημα που προτείνουν είναι, μπορεί και να χρηματοδοτηθεί. Και αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι ναι θα αναλάβουμε εδώ τον ηγετικό ρόλο, ναι θα αναλάβουμε την κυρία πρωτοβουλία αλλά αναμένουμε να ε, μας δείξουν και με σαφή τρόπο οι χώρε χώρες τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν ε, και θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ μας ε, πριν από την Κομπεχάγη. τώρα, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία στον χώρο των οχημάτων, Ναι, ως Προεδρία βρισκόμαστε σε ε, φάση συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και μετά βέβαια είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει τη δική της πρόταση. Όμως εμείς θα ε, κάνουμε όλα τα βήματα από την πλευρά μας για να ξεκινήσει η δουλειά, ε, το νομοθετικό έργο δηλαδή, από την πλευρά της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τον Ιδράργυρο, δεν έχουμε σκοπό να αναλάβουμε νομοθετική δράση σε αυτό το τομέα, όμως έχω ενδιαφέρον για αυτό το τομέα. Υπάρχουν κάποια εθνικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ε, ξεκινήσει και ε, προφανώς ε, προωθούμε ε, την ε, περαιτέρω δουλειά που γίνεται για την κατάργηση του Ιδραρχείου σε εθνικό επίπεδο. Και άρα λοιπόν οι εθνικές συμφωνίες και συνομιλίες θα έχουν εδώ το πλέον σημαντικό ρόλο. Αυτό που θα κάνουμε κατά τη δική μας Προεδρία είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει τις αντίστοιχες πιέσεις. Έχουμε δει τις πρωτοβουλίες αλλά θα πρέπει τώρα να γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι. Έχουμε ήδη συζητήσει με τις ΗΠΑ, με την Κίνα και με άλλους σημαντικούς Τέλος. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική για την βιοπικιλότητα, να πούμε ότι ε, πράγματι και εγώ είμαι απογοητευμένο με το γεγονό ότι δεν έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένου στόχου για το 2010. Όμω θα συνεχίσουμε τώρα τη δουλειά μα σε συνεργασία και με την Ισπανική και με τη Δυτική Προεδρία, ώστε να έχουμε μια σαφή ε, πρόταση για ε, παγκόσμιους στόχους σε ό,τι ε, αφορά τη βιοποικιλότητα αλλά και ταυτόχρονα όπως να θέσουμε και στόχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να τηρήσουμε τα όσα ήδη έχουμε υποσχεθεί αλλά και να κινηθούμε ακόμα παραπέρα ούτω ώστε βέβαια να συμμορφωνόμαστε και με τα όσα έχουμε συμφωνήσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ε, για τις απαντήσεις που δώσατε. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουμε μόνο 35 λεπτά στη διάθεσή μας και 20 ομιλητές. Ε, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα παρακαλέσω όσους, όλους όσους θα λάβουν το λόγο να μιλήσουν μόνο για δύο λεπτά. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε όλα. Δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. κυρία Ρόσπαχ λοιπόν. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά υπευλήθη μία ερώτηση σε σχέση με το τι θα κάνει η Σουηδική Προεδρία στην Κοπενχάγη τον Δεκέμβριο. Ε, και αν κατάλαβα καλά είπε ο κύριος Υπουργό ότι δεν ε, περιμένει να συμφωνηθούν για τη Μαύρη Θάλασσα, για την Μεσόγειο, κάποιοι τους στόχοι δεσμευτικοί. είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ Σουηδίας και Δανίας. Τι, με τις αλληλευτικές συμφωνίες. Είδατε τι έχει γίνει. Δεν έχουν επιτυχθεί συμφωνία για, ε, για, για, την αλληλευτική πολιτική. Επομένως, ε, θα μπορέσετε, είναι, είναι ρεαλιστικό τελικά να συμφωνήσετε με όλες αυτές τις χώρες και τις ε, χώρες που δεν συμφωνούν ε, μεταξύ τους και να κάνετε να συμφωνήσετε κάτι όσον αφορά τη Μεσόγειο αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα. Ε, Κυρία Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας θέσω ερωτήσεις κύριε Υπουργέ. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε όταν μιλήσατε για την ανάγκη μιας οικολογικά αποδοτικής οικονομίας. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, βιώνουμε μία περίοδο κρίσης. Ε, υπάρχουν ταυτόχρονα προγράμματα που πρέπει να, να εντατικοποιηθούν για την ανάκαψη της οικονομίας. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του δημοσίου στην οικονομία της αγοράς θα συνεχίσει να είναι ε, κεντρικός, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου, που είναι σημαντικός για την οικονομία. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να διευκολύνετε την ανάδειξη μεγάλων ε, σχεδίων σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα στις μεταφορές π.χ. Και αν ναι, αυτό αποτελεί κομμάτι της δικής σας ημερήσιας διάταξης. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να τονίσω το ρόλο των πόλεων σήμερα. 80% του πληθυσμού του κόσμου ζει σε 5% της επικράτειας. Δυστυχώς, λόγω της επικουρικότητας, δεν παρεμβαίνουμε στη διαχείριση των πόλεων, ούτε έχουμε σχετική ευρωπαϊκή πολιτική. Το Σεπτέμβριο οργανώνεται μία διάσκεψη με το αντικείμενο αυτό. Τι στόχους έχετε και τι θέλετε να πετύχετε από τα κράτη, τις πόλεις και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω έναν Σουηδό Υπουργό Και είναι σημαντικό το ότι έχετε, η Σουηδία έχει την προεδρία αυτό το εξάμεινο. Μιλήσατε για την σχέση φτωχών πλούσιων χωρών και τη χρηματοδότηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Όπως ξέρετε, υπάρχουν μια σειρά πόρων φορολογικού χαρακτήρα που μπορούν να πάνε απευθείας στην αναπτυξιακή βοήθεια. Μερικές φορές υπάρχουν ωστόσο ορισμένες αντιστάσεις η πρότασή σας, αυτό θέλω να μάθω, πώς θα δομηθεί, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν, δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο έτσι ε, εκκρεμείς υποθε, υποσχέσεις χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχουν νούμερα, συγκεκριμένες υποσχέσεις και θέλω να ξέρω πώς θα πληρώσετε τις προσπάθειες αυτές. Επίσης, θα σας δίνω παράδειγμα. Έχουμε μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εξάγει τις γνώσεις της σε άλλη χώρα. Πώς η επιχείρηση αυτή θα μπορέσει να ενισχυθεί στην προσπάθειά της αυτή. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι ουσιαστικό στον τομέα της χρηματοδότησης. Επίσης, μιλήσατε για την για τη χρήση ε, Τι σημαίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο. Ε, επίσης, μιλήσατε για αυτή την οικολογικά αποδοτική οικονομία. Ωραίο το σχήμα, αλλά τι περιέχει. Στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να ε, μειώσουν τις εκπομπές ε, γιατί μέσω της οικονομίας και άλλοι που πιστεύουν ότι η μείωση θα επιβαρύνει την οικονομία. Τι άποψη έχετε εσείς. Florence, ε, μπορείτε βέβαια να μιλάτε και λιγότερα από δύο λεπτά, τόσο ώστε να προλάβουν σίγουρα όλοι. Έτσι. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε ε, και πρόεδρε του Συμβουλίου, συμφωνώ με τα όλα όσα είπατε μόλις τώρα, αλλά έχω μια ανησυχία, γιατί εγώ είμαι ένας ε, ως μικροεπιχειρηματίας ε, και εγώ ανησυχώ ότι δεν θα έχουμε πλέον ρευστότητα, δεν θα έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Και ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα των τραπεζών δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι στιγμής και εκείνο που προσπαθούν να κάνουν οι περισσότερες τράπεζες είναι να επανέλθουν και πάλι στο status quo, πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε καμία βιώσιμη εδώ χρηματοοικονομική πολιτική. Άρα σας παρακαλώ, εάν όλα αυτά τα οποία συμφωνούμε εδώ και θέλουμε πραγματικά να εφαρμοστούν, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια και θα πρέπει να δεσμεύσουμε ανάλογα τι ε, τράπεζε. Και έχω και εδώ, για παράδειγμα, κάποιες μικρές περιφερειακές τράπεζες ε, μπροστά μου που ξέρω ότι δεν το πράττουν αυτή τη στιγμή. Ε, μετά, σε ό,τι αφορά τους ε, ε έχουμε ε, ε, μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά ε, την εφαρμογή σχετικών διατάξεων. Έχουμε ένα συν για τη Γερμανία 42%, 112% για την Ευστρία και μείον 24% για την Ελβετία. Αυτό το λέω για μερικούς οι οποίοι μπορεί να αναρωτιούνται. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι. Νομίζω πως, μάλλον ελπίζω, πως η σχετική ανησυχία σε ό,τι αφορά τι απτήρες και το όλο το σκάνδαλο, ας το πούμε έτσι, έχει ξεκινήσει μόνο στη Γερμανία, κυρίως στη Νότια Γερμανία και όχι αλλού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσά κύριε Υπουργέ για όσα μα έχετε πει, για όσα μα έχετε απαντήσει στι ερωτήσει. Ε, Εμεί θέλουμε να σα ρωτήσουμε για το τι θα γίνει μέχρι τότε. Ε, και μα χαροποιεί πάρα πολύ το ότι είστε αισιόδοξο για την Κοπενχάγη. Διακόπτη ο πρόεδρος. Ναι, ναι, εσεί, εσεί έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε λέει ο κύριος Παρνιά. Λέγομαι Ζιλ παρνιά και θα ήθελα να σας υποβάλω μια συντομή ερώτηση για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε όσον αφορά τις αντισυκορυφίες. Πώς μπορούμε το συντομότερο τον έχουμε έναν φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα στο, στα στάσινα της κοινότητας. δεν μπορέσουμε να εντάξουμε στην πολιτική μας αυτό το, το κόστος των εκπομπών. Έχουμε από τον ΠΟΕ και από τον ΟΗΕ εκθέσεις όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της ε, ε, την εξέλιξη του της αλλαγής του κλίματος ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες ποσοστώσεις ε, που να μην ε, επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και έτσι να πλήσεται η ανταγωνιστικότητα. Επομένως, να λάβουμε κάποια μέτρα, ούτως ώστε να μην έχουμε ε, εκπομπές, διάχυση, ε, φυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση του, ε, του, του, του γιατί έτσι θα έχουμε 25 εκατομμύρια παραπάνω ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της χρονιάς της φετινής του 2009. Λεπάζω. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας και θέλω να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα κάτι για τα οικονομικά, όπως πολλοί συνάδελφοι τόνισαν, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε κάποια μέτρα οικονομικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Κοπεχάγη, δεν θα αποσπάσουμε αποτελέσματα, μια που τώρα σοβεί η οικονομική κρίση, περιθωρία ελιγμών, ε, τώρα είναι πάρα πολύ μικρά για τις οικονομικές χώρες, δεν τηρούνται υποσχέσει προ τι χώρε του Νότου και επομένω θα πρέπει να δούμε πώ θα βρούμε ένα οικονομικό μηχανισμό να στηρίξουμε τι κινήσει μα. Μα είπατε για κάποιου είδου ε, επιδοτήσεις περιβαλλοντικές, κάτι όμω το οποίο αντιβαίνει προ ε, μια οικονομία περιβαλλοντική, οικονομικά αποδοτική, ε, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδους κονδύλια τα οποία να κατευθύνουν προς αλλού. Δηλαδή να τα ρίξουμε προς την μείωση των εκπομπών των βλαπτικών αερίων στις χώρες του Νότου. Επομένως, τώρα, έτσι και για το πώς θα λειτουργήσει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο μέλλον σε όλο τον κόσμο. Άρα χρειάζεται στενή συνεργασία με αντίστοιχα θεσμικά όργανα για να ζητηθεί μια λύση. Κάτι άλλο τώρα, πιο σύντομο, για αυτή την οδηγία που μας αναφέρατε. Δεν, δεν, δεν, δεν πρόσεξα τι είπατε. Όσον φορά το έδαφος, είναι προτεραιότητα η σχετική οδηγία της, ε, για, για την προεδρία σας. Ευχαριστούμε, Κορίν. Μπελία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τουλάχιστον γιατί δεσμευθήκατε να μεταφέρετε τη μάχη κατά των αλλαγών του κλίματος σαν προτεραιότητα της ε, Σουηδικής Προεδρίας, όπως και τη μάχη για τη μείωση, τη, κατά της μείωσης ε, Σύντομα θα μιλήσω, γιατί πολλά από αυτά που θα τα πω τα είπε η κυρία Λεπάζ. Δεν άκουσα μεταξύ των προτεραιοτήτων σας να αναφέρετε να αναφέρεστε στα οριζόντια κείμενα που αφορούν στην αντιμετώπιση της αλλαγή του κλίματος και της καταπολέμησης της μείωση της βιοπικιλότητα που συζητούνται στο Συμβούλιο Υπουργού εδώ και χρόνια και που έχουν κολλήσει εκεί. Εξηγούμε ποια είναι η θέση σας και ποιες είναι οι προθέσεις σας σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο για το έδαφος, αλλά και την ενσωμάτωση του τρίτου πακέτου της ε, ε, σύμβασης για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Σύντομη και επί του θέματος. Προτείνω και οι άλλοι συνάδελφοι να ε, ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Ο κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την σαφή παρουσίασή σας. Είμαστε, ξέρουμε ότι η Σουηδική Προεδρία συνδέει το περιβάλλον με την ανάπτυξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και χαίρο που δίνεται έμφαση στην ανάγκη, στην ανάγκη αναζήτησης νέων πράσινων λύσεων. Πώς συγκεκριμένα προτίθεστε να καταστήσετε την ανάπτυξη των πράσινων λύσεων σαν πιο δυναμικών λύσεων. Εμείς θα θέλαμε να δούμε εδώ ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ένα πράσινο πρωτάθλημα, ένα πράσινο ευρωπαϊκό κύπελο. Πώς βλέπετε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας σαν βασικό παράγοντα στη διαδικασία αυτή. Okay. <laughs> So, να, να μιλήσω πρόεδρε να μην μιλήσω. Θα είμαι πολύ σύντομος πρόεδρε και Υπουργέ και θα μιλήσω στα Δανέζικα. Πέραν των ευγενειών, να σας πω ότι πραγματικά χαίρο που είστε τόσο αισιόδοξο και φιλόδοξους ε, σε σχέση με το τι θα γίνει στην Κοπενχάγη. Εγώ και άλλοι δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Το είπε η κυρία Μακέβανση. Οι στόχοι που έχουμε που έχουμε παρουσιάσει ε, που έχουν παρουσιάσει οι ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να... Ε, τι, τι, τους στόχους, ε, τι, τι θέλουμε τις, τα συνέδρια αν δεν μπορούμε να, να συμφωνήσουμε επί των στόχων. Και έχω την εξή ερώτηση κύριε Υπουργέ. Όταν συζητάτε τα θέματα αυτά με τους Αμερικανούς, τι σας απαντούν. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι η απάντησή τους είναι δεν κάνετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που λέτε. Μιλάτε, μιλάτε για μείωση 20-30% σε σχέση με το 90% ε, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν απλά να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές. Υπάρχουν όμως και ή εκπομπές από τρίτες χώρες. Εγώ παρακολουθώ τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, διαβάζω τον τύπο και είμαι πεπισμένος ότι χρησιμοποιούν μια σειρά ψευδών επιχειρημάτων που στόχο έχουν μόνο να μας μπλέξουν. Τι απαντάτε σε αυτά. Ε, υπάρχουν ολόκληρα επιστημονικά κείμενα, υπάρχουν οι έρευνες των ε, ειδικών που δεν είναι το που λένε ότι ε, ο στόχος πρέπει να είναι 450 ppm. Ε, τι θα απαντήσουμε σε, αυτά τα, σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Ναι, και σας είπα ότι αναμένουμε ενδιαφέρον να συναντηθούμε, οπότε ε, πραγματικά θα, θα αντισταθώ, θα προσπαθήσω να αντισταθώ στην ε, πρόθεσή μου να απαντήσω σε όλες ε, τις ερωτήσεις ε, λεπτομερώς, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε περαιτέρω επαφή. καταρχήν να πω ότι δεν αναμένω δεσμευτικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά τις διάφορες θαλάσσιες περιοχές. Αναφέρομαι σε στρατηγικές θαλάσσιες και πώς αυτές μπορούν να συνδεθούν με ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τώρα μια οικονομία η οποία θα είναι οικοαποδοτική οικολογικά δηλαδή αποτελεσματική. Εγώ θεωρώ πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει μια δυνατότητα για να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις, για να δημιουργηθούν νέες ε, ευκαιρίε. Ε, και δεν προτείνω εδώ υποχρεωτικά μεγάλα ευρύτερα ευρωπαϊκά project ή έργα αλλά ε, αντίστοιχε προϋποθέσεις μέσω δηλαδή των αντίστοιχων εργαλείων μέσω των κατάλληλων πολιτικών ούτω ώστε να αναπτυχθούν σχετικέ τεχνολογίε, να δοθούν τα ερεθίσματα για την δημιουργία βιώσιμων πόλεων περιβαλλοντικά βιώσιμων πόλεων και όλα αυτά θα μπορούσαν να ε, μπουν μέσα στον ε, διάλογο που θα γίνει κατά τη διάρκεια της δικής μας ε, Προεδρία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα χρηματοδότησης και τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τις εγκληματικές μεταβολές. Προφανώς, εάν δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν υπάρχει συμφωνία. Σύμφωνοι, αλλά αυτό που υπογραμμίζω ξανά και ξανά ότι πληρώνουμε για κάτι. Εάν λοιπόν αυτές ε, μειώσεις ε, των εκπομπών ε, δεν εφαρμοστούν στην πράξη, τότε δεν θα πληρώσουμε τι αυτές. Δηλαδή, εάν δεν υπάρξουν μειώσεις των εκπομπών, δεν θα καταβληθούν κονδύλια. Άρα λοιπόν ζητούμε από τις χώρες να ε, θέσουν επιτάπητο στα δικά του σχέδια για τη μείωση των εκπομπών, ώστε να είμαστε βέβαιοι και εμεί από τη δική μα πλευρά ότι καταβάλουμε κονδύλια για δράσει οι οποίε λαμβάνουν χώρα. Και γι' αυτό λέμε ότι όσα θα πρέπει ε, να γίνουν εδώ θα πρέπει να είναι και βιώσιμα από χρηματοδοτική άποψη και γι' αυτό χρειαζόμαστε και ε, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ιδιωτική χρηματοδότηση και ε, συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε μόνο αυτέ τι αποφάσει, αλλά χρειαζόμαστε και του κατάλληλου μηχανισμού για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτού του στόχου και γι' αυτό θεωρούμε πω είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτού του μηχανισμού σε ό,τι αφορά την προσαρμογή και την μεταφορά της ε, τεχνολογίας, ε, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη δημιουργία αντίστοιχων δυνατοτήτων στις ε, πιο φτωχές χώρες. Εκεί χρειάζονται τα κονδύλια. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών χρειάζονται αυτά τα κονδύλια και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το CDM. Είναι προφανές ότι το σημαντικότερο κομμάτι θα πρέπει να εφαρμοστεί να υλοποιηθεί εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά όμω είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε στις ΗΠΑ και σύντομα θα έχω να, δυνατόν να προβώ σε διάλογο με την νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Έχω ήδη συναντηθεί με τους ε, αρμόδιους ε, του εν λόγω κόμματος ε, αρκετές φορές και θα το υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι θα πρέπει η εθνική δράση και είναι σωστό η εθνική δράση να συμπληρωθεί από διεθνή δράση. Γιατί κάτι τέτοιο μπορεί ακριβώ να δώσει το ανακτήριο λάκτισμα για την ανάληψη πρωτοβουλειών από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών. Άρα λοιπόν το CDM δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι ε, κάτι το υπερβολικά δύσκολο, ότι θέτουμε υπερβολικά ψηλά το πύχη, μπορεί να θεωρηθεί ως ε, το έναυσμα για να ξεκινήσουν αντίστοιχε πρωτοβουλίε σε άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην αρχή, αλλά θα πρέπει να οδηγηθούν τελικά στην ε, τελική κατάργηση. Ε, νομίζω πως αναφέρθηκα στα κυριότερα ζητήματα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα εδάφη. Ε, είδαμε ότι μια σειρά από προεδρίες έχουν καταβάλει προσπάθειες εδώ. Η τσεχική προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά ε, όταν προσπάθησε να βρει μια λύση και νομίζω πως ε, τώρα έφτασε η ώρα να αναλογιστούμε σε πολιτικό επίπεδο το πώς θα προχωρήσουμε μελλοντικά, ούτως ώστε ένα συγκεκριμένο επόμενο βήμα να γίνει κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα όσα είπε ο Καρχάλης ε, Φλόγανς, ε, και εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ε, προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν χρειαζόμαστε μία σειρά από δύσκολου κανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συγκεκριμένε τοπικέ λύσει για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και τέλος, ναι, πολλές ανεπτυγμένες χώρες ε, βρίσκονται πολύ πιο πίσω ή κάνουν πολύ λιγότερα σε σχέση με τα όσα θα πρέπει να κάνουν ώστε να επιτύχουμε τη μείωση ε, των δύο βαθμών. Οπότε η δική μου στάση είναι ότι ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξο ω προ το ότι αυτό θα επιτευχθεί. Απλά είμαι αισιόδοξο ως προς το ότι εδώ υπάρχει ανάγκη ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλία και εδώ ε, λέω πως η Ευρώπη από κοινού δηλαδή ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, ε, η πολιτική γενικά και το ευρύ κοινό στις χώρες μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, όλες αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να έχουν αυτό το ρόλο αφού έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση και να μπορέσουμε ακριβώς να κινητοποιήσουμε άλλες χώρες. Αναμένουμε περισσότερα από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Φυσικά, αναμένουμε περισσότερα και από άλλες ε, χώρες. Αλλά θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο και να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτόν τον ρόλο. Δεν αποτελεί εγγύηση, αλλά τουλάχιστον εκ των υστέρων θα μπορούμε να πούμε πως κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένας σύντομος τρίτος γύρος τώρα ο καθένα από ένα λεπτό. Κυρία Κουτήρες Κορτίνε. Oh. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Γιατί έχουν ε, δύο θέματα τα οποία με απασχολούν. Πρώτα πρώτα να σας ε, πω κάτι το οποίο μπορεί να σας φαίνεται οδυνηρό, επώδυνο, αλλά δεν υπάρχουν ηγέτες χωρίς οπαδούς. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, ό,τι περιεχόμενο και να δίνουμε ε, στην πρωτοπορία, στην έννοια πρωτοπορία για το, για το ε, κλίμα, για τον αγώνα αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι θεματικό και εντυπωσιακό. Όμω χρειάζονται κάποια, κάποια μέτρα, τόσο ώστε να ακολουθήσουν κάποιοι του πρωτοπόρου και μέτρα τέτοια δεν έχουμε λάβει. Εμένα πάρα πολύ με, με απασχολεί το πώς συνολικά βλέπουμε το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το βλέπουμε πιο σφαιρικά, που δεν το βλέπουμε τώρα, ε, σε σχέση δηλαδή ε, με το τι γίνεται με τη γεωργία και τις εκπομπές. Είναι κάτι το οποίο δεν βρήκε συνέχεια, επομένως χρειάζεται κάποιο είδους περιφερειακή εφαρμογή των μέτρων για το κλίμα. Αλλιώς ε, δεν πρόκειται οι, οι περιφέρειες να έχουν κάτι για να μπορέσουν να αξιολογήσουν το ρόλο τους. Άρα χρειάζεται συνολικά να το δούμε το ζήτημα. Ε, θα πρέπει επιστημονικά να δούμε το θέμα και όσον αφορά τη σύλληψη των μέτρων και όσον αφορά την εφαρμογή του. Τώρα μια ερωτησούλα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εμεί έχουμε την Προεδρία αργότερα, Εμεί η Ισπανία και αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι το ότι δεν αναφέρεστε καθόλου σε κάποια μεσογειακή πολιτική όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο. Γιατί έχουμε κάποιε αναδυσσόμενε χώρε σαν την Τουρκία, σαν την Αίγυπτο, σαν το Μαρόκο που έχουν τρομερή αύξηση του πληθυσμού. Ε, και επομένως γι' αυτό με εκπλήσει το ότι δεν έχετε μια πολιτική μεσογειακή για το περιβάλλον. Έχετε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Βιτόριο Πρώτη, έχετε ένα λεπτό και Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Βασίζομαι στο γεγονός ότι ήδη μιλήσαμε κάπω για τα προβλήματα αυτά Χθε χάρη στην ευγένεια και την διαθεσιμότητα που δείξατε. Πρώτη παρατήρηση πιστεύω ότι στις ε, προτάσεις της Ευρώπης λείπει μία ρήτρα δικαιοσύνης, ευθυδικίας μάλλον για να έχουμε τη συνένεση των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεύτερον, με βάση το σλόγγαν ένα άτομο, ένα δωρεάν, μία δωρεάν, ένα δωρεάν δικαίωμα εκπομπής. Αυτό είναι βασικό. Άλλο ζήτημα τα τροπικά δάση. Ε, η καταστροφή τους συμβάλλει κατά 20% στις εκπομπές. Με τα μέσα που έχουμε μπορεί να μετατραπούν στον ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο αντιμετώπισης των εκπομπών. Εξού και το πρόβλημα να έχουμε ε, διαγωνισμούς για να πετύχουμε στην, την ε, εκμετάλλευση των δυνατών αυτών. Τρίτον, η διατήρηση του περιβάλλοντος του, χώρου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εκμετάλλευσης των δασικών και γεωργικών υπολοιμάτων. Και αυτό απαιτεί κοινή δράση για να συνεργαστούν οι διάφοροι τομείς στο σημείο αυτό. Και αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωσέ Μανουέλ, Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Καλημέρα. Σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε περισσότερο το θέμα της οικολογικής αποδοτικότητας, το θέμα της οικολογικής αποδοτικότητας, το θέμα του νερού. Σας υπενθυμίζω ότι ε, κάποιοι δημόσιοι φορείς ε, παροχής ύδατος έχουν σε απώλειες 40% και πάνω. Πιστεύω ότι εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να θέσουμε στόχους για να μειώσουμε τις απώλειες αυτές και να πετύχουμε τους στόχους της μείωσης. Και να τους θεσπίσουμε βέβαια. Πέραν αυτού, την οικολογικό, στο θέμα της οικολογικής αποδοτικότητας μήπως θα έπρεπε να θέσουμε ένα στόχο στην ε, μείωση της ε, υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος. ό,τι αφορά τώρα τις παράκτιες περιοχές, το πρόγραμμα της, της Προεδρίας ε, μιλά για την προστασία του ενάλλειου περιβάλλοντος και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ περιοχών και περιφερειών. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε κάπως περισσότερο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τις παράκτιες περιοχές. Και το ρωτώ αυτό λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές αλλαγές που θα προκύψουν λόγω του, της αλλαγής του κλίματος στις περιοχές αυτές. Μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε δράσεις μεταξύ των κρατών μελών για να ή να υπάρξει ας πούμε ένας ευρωπαϊκός χάρτης ε, παραθαλάσσιων περιοχών που αντιμετωπίζουν κινδύνους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Υπουργέ να επανέλθω στο θέμα των ε, χρηματοοικονομικών μέτρων. Είναι το πρώτο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσουμε για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία στην Κοπενχάγη. Ήδη αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποιος μηχανισμός για περιβαλλοντική ανάπτυξη και λοιπά. Και θεωρώ ότι πέραν όλων των άλλων χρειάζεται, χρειάζονται κάποια μέτρα στήριξη. Έχουμε αυτή τη δέσμη μέτρων που ανέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενέργεια και για το περιβάλλον και μιλήσαμε για αυτό το, το, το Ταμείο Προσαρμογής που θεωρώ ότι θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο για να δούμε πώς αυτό το Ταμείο Προσαρμογής θα χρηματοδοτηθεί, πώς θα υποστηριχθεί οικονομικά. συγκεκριμένα να δούμε τι θα γίνει με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την, την, ε, την ευθύνη των Αφρικανικών χωρών με τις χώρες της λεγόμενης BRIC. Voorzitter, en ik wil de minister Kalgreen hartelijk danken voor zijn bijdrage tot zover. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για όσα μας είπε μέχρι τώρα. Μου δημιουργεί εμπιστοσύνη για το τι θα πετύχει η, προεδρία, η Σουηδική Προεδρία το επόμενο, τους επόμενους μήνες. Τονίζεται τη σημασία της Κοπενχάγης. Πραγματικά ε, το κλίμα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταχύτατα και πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η προοπτική να γίνουν μη αναστρέψιμες και μη ελέγξιμες οι αλλαγές στο κλίμα, πρέπει να μας οδηγήσουν σε ακόμα ταχύτερη δράση. Ακόμα πιο επικίνδυνο όμως είναι το θέμα της βιοπικιλότητας, το οποίο είναι ήδη, οι αλλαγές, στο, όπου οι αλλαγές έχουν ήδη γίνει ανέλεγκτες. Η βιοπικιλότητα χρειάζεται ε, να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα, να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο και ίσως γι' αυτό η Προεδρία να ε, μπορεί να παίξει ένα σωστό ρόλο στο θέμα αυτό. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι την άλλη εβδομάδα θα, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για την συνάντηση της επόμενης εβδομάδας υψηλού επίπεδου αφορά μόνο τη βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και εκτός, γιατί πρέπει να είμαστε, να πούμε την αλήθεια. Η καταστροφή της βιοπικιλότητας στις φτωχές περιοχές του κόσμου είναι ακόμα πιο ε, πήγουσα από ό,τι και σε εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, κάνουμε πολύ, ε, γίνεται πολλή δουλειά από τη δική μας πλευρά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε ε, την, ε, την αυτό το 20% εάν αυτό επαρκεί για να επιτύχουμε τα όσα θέλουμε. Ίσως να πρέπει να φτάμε στο 40% Ίσως θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν το 40% και ε, από εκεί και μετά αφού θέσουμε το 40% να αναζητήσουμε την υποστήριξη ε, στο, ε, στο βαθμό που μπορούμε και τότε θα έχουμε και τη μεγαλύτερη αγορά σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, σε ό,τι αφορά την οικολογία, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος και νομίζω πως μόνο τότε θα ανοιχτούν και είπα γιατί τότε θα δημιουργηθούν πραγματικές επενδυτικές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή οι αναπτυσσόμενε χώρε οι οποίε ουσιαστικά ε, ε, ε, υπομένουν το κόστος λόγω των δικών μας εκπομπών θα πρέπει πραγματική, να λάβουν πραγματική υποστήριξη. Άρα λοιπόν θέλουμε φιλόδοξου, πιο φιλόδοξου στόχους, πολύ συγκεκριμένα στόχου στόχους και πολύ συγκεκριμένη και χρηματοδοτική στήριξη. Τότε νομίζω πω όλοι θα συμφωνήσουν ο λόγο ε, σε εσά ε, και πάλι κύριε Υπουργέ. Δυστυχώ και ε, ζητώ συγγνώμη, 8 συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο. Ε, Όμω θα σα δώσουμε τώρα το λόγο για να απαντήσετε. Έτσι καλώ θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν ξανά μαζί σα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τα έντατα και ε, τη συζήτηση ως προς τα ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα ήθελα να πω πως υπάρχει εδώ ε, ανάγκη εξέβρεσης λύσεων για τις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Έχει γίνει πλέον από γεωγραφική άποψη τόσο μεγάλη η Ευρώπη, ούτως ώστε δεν μπορούμε να βρούμε μια έννοια λύση για το σύνολό της. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, επιμέρους λύσεις και γι' αυτό βέβαια ε, βασιζόμαστε και σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία που θα κάνουμε με την Ισπανία σε ό,τι αφορά ε, την Ισπανία την, συγγνώμη, τη Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τροπικά δάση, πράγματι συμφωνώ μαζί σα, κύριε Πρότυπο, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό ε, ζήτημα στο πλαίσιο τη ε, διάσκεψη που θα γίνει. Η δική μα ε, θέση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφή ότι δηλαδή θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά το ίμιση ρωτώ με αυτό των δασών. και να έχουμε ένα τομέα ο οποίος εδώ θα μπορεί να είναι ανοιχτός και για την ε, συγχρηματοδότηση και ταυτόχρονα και για την συμμετοχή της ε, ιδιωτικής ε, πρωτοβουλίας, ώστε να επιτύχουμε τη δική μας μείωση εκπομπών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε σαφή ενεργητική δράση σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα και τη μείωση τη καταστροφή αυτών των δασών με ε, μια συμφωνία η οποία θα επιτευχθεί στη Κοπεχάγη. Και εδώ ευθυγραμμίζομαι λοιπόν με τις δικέ σας ε, προσδοκίε, του δικού σας στόχου, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τώρα και πάλι τα ύδατα και την ε, ανάγκη επίτευξη παράκτιων ε, λύσεων. Δηλαδή, σε παράκτητες περιοχές, ε, ναι, είναι πολύ σοφό να ε, εξετάσουμε το πού ακριβώς βρίσκεται εδώ η ζήτηση για τέτοιες λύσεις, ειδικότερα στην Νότια Ευρώπη. Αλλά και εδώ πάλι διαφαίνεται ακριβώς η ανάγκη εξέβρεσης διαφορετικών λύσεων για τις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης και γι' αυτό αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα γίνει για τη Μεσόγειο και τη συνεργασία που θα έχουμε με την περιοχή της ε, Μεσογείου αλλά και την ε, μελέτη που θα λάβουμε σε σχέση με αυτήν κατά την συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θα βασιζόμαστε και σε σχέση με τη Μεσόγειο ε, σε περιφερειακές πολιτικές και η Βαλτική θάλασσα για παράδειγμα αποτελεί ένα στοιχείο στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής δηλαδή των περιφερειακών λύσεων. Τώρα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή adaptation. Ε, η χρηματοδότηση της προσαρμογής ε, θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες τουλάχιστον για μένα. Γιατί πραγματικά αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό για τις πλέον φτωχές και πλέον ευπαθείς χώρες. Και γι' αυτό κατά κατά τελευταία διάσκεψη εργάστηκα προς αυτό το στόχο ιδιαίτερα. Δηλαδή να δοθούν οι σωστές προϋποθέσεις για αυτά τα ταμεία προσαρμογής ούτω ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Ε, και με την Κοπεχάγη θεωρούμε πως ε, αυτά τα ταμεία προσαρμογή θα μπορέσουν να είναι σε θέση να σηματοδοτήσουν συγκεκριμένα πλέον έργα, συγκεκριμένα project. Θα πρέπει βέβαια να αναβαθμίσουμε και τα όσα θα χρηματοδοτηθούν και μέσω του Ταμείου ε, Προσαρμογής αλλά και μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης. Και εδώ το σημαντικό είναι πως οι αναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει οι ίδιες να μπορούν να έχουν λόγο ω προ το πώ οργανώνονται όλα αυτά, δηλαδή το τι σημαίνει σε επίπεδο διακυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, βιοπικιλότητα, θα ήθελα να συνδέσω αυτό το ζήτημα ε, σε σχέση με τα όσα είπαμε προηγουμένω σε σχέση με τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Η βιοπικιλότητα λοιπόν δεν ε, αφορά μόνο την επίτευξη των όσων είναι αναγκαία ε, από επιστημονική άποψη, αλλά θα πρέπει να ε, επιτευχθούν τα όσα πρέπει να επιτευχθούν και από πλευρά ισότητα. Δηλαδή, κατά τη δική μα ε, Προεδρία, η βασική προτεραιότητα θα είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το ABS, δηλαδή το δικαίωμα των αντισώμενων χωρών να έχουν κάποιο όφελος από τα όσα εμείς καταφέρουμε να αντλήσουμε από τους ε, γενετικούς ε, πόρους ε, και τη γενετική ποικιλότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τέτοιου είδους στόχους πριν από την πνοή της CBD το επόμενο χρόνο. Ναι, σε ό,τι αφορά το κλίμα, προφανώς όπως είπατε και εσείς συνάδελφοι χρειαζόμαστε έναν Al εγωγικών και για μας και ε, με αυτή την έννοια θίξαμε και τις ανάγκες μιας ε, πλατφόρμας ε, και γι' αυτό είπαμε πως θα πρέπει να εκπονηθεί και εν λόγω μελέτη η οποία θα ερευνεί ακριβώς τη σχέση μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και βιοποικιλότητας και ελπίζουμε πως και το Κοινοβούλιο και ε, του Συμβουλίου θα ενδιαφέρονται πάρα ε, πολύ για αυτόν ε, τον τομέα στο μέλλον γιατί δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με απλά κάποια πολύ σημαντικά λουλούδια ή κάποια πολύ σημαντικά φυτά και κάποια πολύ σημαντικά εριζόν αλλά έχουμε πραγματικά να κάνουμε με ένα τομέα που έχει σαφέστατες επιπτώσει στον τομέα της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές μεταβολές καταρχήν δεν ε, εξαιρούμε εκ των προτέρων ε, τυχόν δράσεις ή αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα σύνορα. προφανώς και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε να έχουμε και πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες, δηλαδή για πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Εάν αποτύχουμε, τότε θα δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά ε, πάση περιπτώσει ε, σε, ε, πάντα είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και δεν θα θέλαμε προσαρμογή σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, φόρο ο οποίος τυχόν θα καταβάλλεται στα σύνορα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ε, καταρχήν και αναμένουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη Κοπενχάγη. Ο δικός μας στόχος βρίσκεται στο 30%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τη βούλησή της να μειώσει κατά 30% τις δικές εκπομπές εάν και τα άλλα μέρη, δηλαδή άλλες χώρες, συμφωνήσουν ότι θα πράξουν κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι ε, η θέση του Κοινοβουλίου και εγώ συγκλίνω εδώ με την άποψή του. Ε, δεν είναι δηλαδή δική μου αυτή η άποψη. Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε. Το Συμβούλιο θα κληθεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, τα ίδια τα κράτη-μέλη θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ σημαντικό στην περαιτέρω δουλειά που θα γίνει και ελπίζω πως ε, θα έχω τη δυνατότητα να ακούσω για μία ακόμα φορά τις απόψεις σας και να διευρύνω τον διάλογο μεταξύ μας και η δική σας ε, συμβολή θα είναι ε, πολύ σημαντική την προώθηση αυτής της περιβολωτικής ατζέντας την οποία συζητήσαμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας, σας ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Λάινο και σας αναμένω με ενδιαφέρον βέβαια και τη συμμετοχή σας στις προχώμενες διασκέψεις στους επόμενους μήνες. Αγαπητέ Υπουργέ, κύριε Αντρέα Κάγκρεν, πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε το μεγάλο ενδιαφέρον από τη δική σα ε, πλευρά και από την πλευρά τη Σουηδική ε, Προεδρία γενικότερα. Ζητώ και πάλι συγγνώμη από του 8 συναδέλφου που δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο. Θα έχουν ε, την προτεραιότητα στην επόμενη φορά που θα γίνει με τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Και συνεχίζουμε τώρα κατευθείαν με τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Γκίντα Φαχόη. Uh,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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξή μα. Σα ε, παρακαλώ, λάβετε θέσει. Ε, Όποιο δεν θέλει να παραστεί στη συνεδρίαση, να εξέλθει από την αίθουσα. Όσοι θα συμμετάσχετε, καθίστε, τόσο ώστε να επανέλθουμε λίγο στην, στο πνεύμα εδώ των εργασιών μας. Αντιλαμβάνομαι πως υπήρξε έτσι αυτό το μεγάλο διάλειμμα, το καλοκαιρινό και υπάρχουν πολλά που θέλετε να συζητήσετε, αλλά εάν υπάρχουν άλλοι με άλλες ανηλυμένε υποχρεώσεις που θέλουν να συζητήσουν, έχουμε ένα μεγάλο κτίριο στη διάθεσή μας, οπότε μπορείτε να συζητήσετε όλα αυτά εκτός εθούσης. Ωραία. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής ε, διάταξης ε, έχω λοιπόν την τιμή να ε, καλωσορίσω σήμερα εδώ τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ε, τον κύριο Γκίντα Φαχόγγιν, στην Επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν, ευθύ εξ αρχής με την έναρξη της νέας βουλευτικής θητείας, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Φαχόγγιν το φαρμακευτικό πακέτο. Κύριε Φαχόγγεν, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην Επιτροπή μας και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε το τι θα γίνει ε, μελλοντικά σε αυτό το τομέα ε, με το νέο πλέον ε, κοινοβούλιο και βέβαια την Επιτροπή η οποία σύντομα και αυτή θα ανασταθεί. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Ε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμε κύριε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για την, ε, πρόεδρε, για την εκλογή σας ε, σε αυτό το αξίωμα του Προέδρου λοιπόν, αυτής της σημαντικής επιτροπής του Κοινοβουλίου και σας ε, συγχαίρω βέβαια όλους για την εκλογή σας ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δική μου θητεία δεν ξέρω κατά πόσο θα διαρκέσει όσο και η δική σας. Αυτό βέβαια εξαρτάται σε ένα βαθμό από εσά. Αλλά σας διαβεβαιώ πως ε, ε, μέχρι και την τελευταία ημέρα θα, ε, πληρώσω, θα τηρώ στο ακέραιο τις δικές μου υποχρεώσεις και θα είμαι στη διάθεσή σας έως και την τελευταία ημέρα που εγώ θα κατέχω το δικό μου αξίωμα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια σημεία, σε κάποιους ε, φακέλους, σε κάποια θέματα τα οποία ήδη έχετε ε, εξετάσει. Καταρχήν ε, να σας πω πως η πρώτη συνάντηση που κάνουμε κοινοβουλευτική επιτροπή στο νέο κοινοβούλιο είναι με τη δική σας επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθώς ε, θεωρώ πως θα επιτύχουμε ε, αυτή την υπέρβαση, την επιτυχία σε ό,τι αφορά μια ε, νέα οικονομική μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μια πολιτική οικονομία η οποία κατά κύριο λόγο θα εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην βιωσιμότητα, στην αεφορία. Ε, και σας το λέω αυτό εμφατικά, κατά κύριο λόγο θα εστιάσουμε σε αυτό, εν ώψη και της ε, κρίσης η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 12 ε, μήνες και ε, εξετάζοντας τα όσα είδαμε και κατά την προηγούμενη βουλευτική θητεία. Ε, θα κάνω λοιπόν ένα σχόλιο το οποίο μπορείτε να εκλάβετε και ως παράκληση από την πλευρά μου. Αυτό το τεράστιο καθήκον το οποίο έχουμε μπροστά μας θα έχει επιπτώσεις ε, για ε, ε, ολόκληρη τη ζωή μας. Όχι δηλαδή, θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο για τον τρόπο παραγωγής μας, αλλά και για τον τρόπο κατανάλωσής μας. Δηλαδή θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και να εγκαταλείψουμε λίγο τα ιδεολογικά χαρακόμματα τα οποία είχαμε καταλάβει στο παρελθόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να μην διατηρήσουμε παλιά, παλιές εικόνες, ε, παλιούς τρόπους σκέψης σε ό,τι αφορά τους εχθρούς που έχουμε για παράδειγμα. Ε, δηλαδή να λέμε για παράδειγμα η βιομηχανία είναι η κακή. Η, αυτή είναι η κακή, αυτοί θέλουν το κακό μας. Η επιστήμη έχει ένα διφορούμενο ρόλο, δηλαδή μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κακή, ανάλογα, και εμείς είμαστε οι καλοί. Κάτι τέτοιο δεν μας βοηθάει. Εκείνο που μας βοηθάει είναι να επιτύχουμε μία κοινή αντίληψη ως προς το ότι χρειαζόμαστε τα όσα μας προσφέρει τόσο η επιστήμη όσο και η βιομηχανία για να επιτύχουμε το κατάλληλο ισοζύγιο εδώ. Και σας το λέω αυτό όχι μόνο επειδή είμαι πεπισμένος πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε μακροπρόθεσμα στο δικό μας πλανήτη, αλλά και επειδή χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο ούτως ώστε η Ευρώπη να, αποτελέσει, να, να, να έχει μάλλον ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον η Ευρώπη. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο που πλέον θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ε, την ε, διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στις σε οικονομία. Ε, πραγματικά είμαι σήμερα ακόμα ε, πιο πεπισμένο ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η λήψη υπόψη περιβαλλοντικών ε, παραμέτρων δεν αποτελεί απλά ένα ζήτημα, αν θέλετε, ένα επιπλέον παράγοντα κόστους, ο οποίος μπορεί να ληφθεί υπόψη όταν έχουμε καλύψει ήδη όλα τα υπόλοιπα ε, προβλήματα και όλους τους παράγοντες ε, κόστους. Όχι, ευθύς εξ αρχής στον προϋπολογισμό, αν θέλετε, ε, στους υπολογισμούς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και αυτός ο παράγοντας, ο περιβαλλοντικός παράγοντας. Εάν λοιπόν αντιληφθούμε ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει τόσο από τα επιστημονικά ιδρύματα όσο και από τις εξελίξεις που έχουμε στην τεχνολογία και όσο και από την πλευρά της βιομηχανίας έχουμε βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση, κατέχουμε ηγετική θέση εδώ. Και άρα λοιπόν η κοινή μας ευθύνη θα πρέπει να είναι να αξιοποιήσουμε ακριβώς αυτή την ηγετική θέση, αυτή την ε, πλεονεκτική θέση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν θα μπορέσω να κάνω πολλά βέβαια στους υπολοιπούς επόμενους μήνες που θα κατέχω αυτό το αξίωμα, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ το εν λόγω μήνυμα ε, να το μεταδώσω και στον συνάδελφο που θα αναλάβει αυτή την ε, θέση. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η οποία χτύπησε την παγκόσμια οικονομία κίνδυνος του να ξεχάσουμε μαθήματα που είχαμε μάθει στο παρελθόν ε, δεν επαληθεύτηκε τελικά. Άρα δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για τη διαχείριση της κρίσης είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει να ε, συνεπιφέρουν τον κίνδυνο του να ε, αμβλύνουμε ε, τους μακροπρόθεσμους ε, στόχους μας. Έγιναν λοιπόν κάποιες πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να μειώσουμε τις προηγούμενες προσπάθειες που είχαμε κάνει. Ε, αντιθέτως, εκείνο που είδα εγώ είναι ότι υπάρχει μια ε, ευρεία συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή ο οικολογικός προσανατολισμός και η ε, χρηστή διαχείριση των πόρων αποτελούν και θα πρέπει να αποτελέσουν ε, εργαλεία ε, διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Και εμείς από την πλευρά μας είπαμε με πολύ σαφή τρόπο στις επιχειρήσεις μας, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ότι ε, ε, θα πρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση η οποία χρειάζεται βέβαια και ε, περαιτέρω επενδύσεις. Και προφανώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αντίστοιχα αυτός ο αναπροσανατολισμός, ο οικολογικός αναπροσανατολισμός. Αυτό ε, λοιπόν ήταν το πολιτικό μήνυμα το οποίο μπορώ εγώ να εκφράσω ε, και το οποίο έχω αποκομίσει από τα ε, πέντε χρόνια της προϋπηρεσίας μου εδώ. Ε, επιτρέψτε μου τώρα να περάσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Ε, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης βουλευτικής θητείας Ακούσατε βέβαια για τα όσα είχαν συζητηθεί σε ό,τι αφορά το φαρμακευτικό πακέτο και τη στρατηγική για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα ε, με τρεις ε, νομοθετικές πράξεις οι οποίες σχετίζονται με την εποπτεία των ε, συσκευασμάτων, την προστασία τους από απομιμήσεις και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, και επίπεδο, δηλαδή την πληροφορία, την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά στήματα. Ε, ε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν γίνει λοιπόν πριν από τη λήξη τη βουλευτική ε, θητεία του προηγούμενου δηλαδή κοινοβουλίου, ε, επιτεύχθηκαν πολύ σημαντικά πολύ σημαντική πρόοδο ε, σε ό,τι αφορά τόσο τον τομέα τη εποπτεία όσο και τη ε, προστασία των φαρμάκων από απομιμήσει. και δεν ε, φοβούμε εδώ πώ θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Εκφράζω λοιπόν την αισιοδοξία μου ότι θα κινηθούμε γρήγορα σε αυτού του τομεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία γνωρίζει σε τι θα πρέπει να προσαρμοστεί. Και στου δύο λοιπόν αυτού τομεί, και στον χώρο τη εποπτεία και στον χώρο τη προστασία από απομιμήσει, δεν θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι να προκύψουν κάποιες ε, καταστροφές για να κάνουμε κάτι και αν δεν κάναμε κάτι θα προέκυπταν σίγουρα κάποιες καταστροφές. Θα πρέπει λοιπόν να κινούμαστε προληπτικά και γι' αυτό ακριβώς έχει φτάσει το σωστό χρονικό σημείο για να αναλάβουμε δράση σε αυτούς τους τομείς. Το δύσκολο ζήτημα είναι η ενημέρωση των ασθενών. Ο τρίτος τομέας. Και γνωρίζω πως είναι και ένα λεπτό ζήτημα. Εγώ θα πρέπει να πω πως ε, είμαι πλέον ε, πιο πεπισμένος από κάθε άλλη φορά πως είναι απολύτως απαραίτητο προς τον συμφέρον των ασθενών να φτάσουμε σε νομική σαφήνεια εδώ. Η πρόταση της Επιτροπής δεν βασίζεται στα συμφέροντα της ε, φαρμακοβιομηχανίας και οτιδήποτε άλλο. Ε, βασιζόμαστε εδώ και προσανατολιζόμαστε προς το συμφέρον των ασθενών και θα πρέπει να σας πω πραγματικά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ γιατί στον τομέα της υγείας. Όλοι όσοι ε, δραστηριοποιούνται εδώ επαγγελματικά, όσοι δηλαδή εδώ έχουν ως στόχο την, ε, το κέρδος λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και τελικά όλοι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν το όφελος αν θέλετε, όσοι δηλαδή εκείνοι ε, οι οποίοι τελικά είναι εκείνοι για τους οποίους παράγονται αυτά τα σκευάσματα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Δεν θέλω εδώ να σας ε, ε εκφράσω κάτι συναισθηματικά ε, αλλά ίσως να ε, έχετε βιώσει κάτι αντίστοιχο στη δική σας ε, οικογένεια, ε, δηλαδή του να έχει ασθενήσει κάποιος βαριά και όλοι, δηλαδή οι συγγενείς, οι φίλοι προσπαθούν και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δουν κατά πόσο υπάρχει μια άλλη αποτελεσματική θεραπεία. Και όποιος βρεθεί σε αυτή την κατάσταση θα έχει μια αντίστοιχη στάση, δηλαδή δεν θα μπορεί να αντιληφθεί γιατί θα πρέπει τέτοιου είδους πληροφορίες να μην είναι προσβάσιμες. Γιατί να μην μπορούν να είναι αυτές οι πληροφορίες ε, διαθέσιμες και προς επαλήθευση ω προς την ε, εγκυρατητά τους. Ε, είναι λοιπόν απαραίτητο να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Καταρχήν έχουμε και εδώ και κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Έχουμε γύρανση του πληθυσμού. 15% του πληθυσμού μας είναι άνω των 60 ετών και ε, αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ο τομέας της ε, δημόσιας υγείας γίνεται όλο και πιο ε, σημαντικός και η ανάγκη σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Άρα λοιπόν η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες ταυτόχρονα αυξάνεται βέβαια τρομακτικά. Ε, και ε, μέσα στα 10 χρόνια είδαμε πολύ, πολύ σημαντικές αλλαγές και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά θα εξελιχθούν ακόμα περαιτέρω. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το υπόβαθρο θα πρέπει να κάνουμε ένα ελεγχόμενο, ένα προσεκτικό βήμα και αυτό ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλωστε είναι απαραίτητο και με βάση την ομολογία, τη μέχρι τώρα ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το να χαρακτηρίζει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ τη ενημέρωση και τη διαφήμιση. Ε, δηλαδή το κύριο μέρο εδώ τη ομολογία προέρχεται από το ΔΕΚ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ε, πράγμα το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως επαρκεί. Κάτι ακόμα να πω. Και εγώ θεωρώ πως ε, στο πλαίσιο της φαρμακοβιομηχανίας και των συναφών ε, τομέων υπάρχουν κάποιες πρακτικές ε, προώθησης των πολίσεων οι οποίες πραγματικά είναι απαράδεκτες. Δεν είμαστε αφελείς. Ασφαλώς γνωρίζουμε ποια τεχνάσματα χρησιμοποιεί για να καταστρατηγήσει την απαγόρευση της διαφήμισης της φαρμακοβιομηχανία. Για παράδειγμα, πώς το καταστρατηγεί τόσο σε έντυπα μέσα, όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα, Υπάρχουν κάποιες εδώ, κάποια άρθρα τα οποία δημοσιεύονται και κάποιες ενημερώσεις, ε, οι οποίες όμως τελικά, σε τελική ανάλυση, προέρχονται από την ίδια τη φαρμακομηχανία. Χωρίς βέβαια στον καταναλωτή, σε εκείνον που διαβάζει αυτό το άρθρο, να δίνεται αυτή η διευκρίνηση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θέτει ως προϋπόθεση ότι η ενημέρωση, η πληροφορία που δίνεται στο, στους ασθενείς θα πρέπει να ε, συνδέονται άμεσα με ένα κώδικα δεοντολογίας, ένα code of conduct, ούτως ώστε οι εν λόγω ε, πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται πάντα σε αυτή την γκρίζα ζώνη και τις οποίες βλέπουμε τόσο συχνά να καταργηθούν παντελώς. Έτσι λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο θα υπάρξουν διαθέσιμες περισσότερες και πιο έγκυρες πληροφορίες για τους ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα οι ασθενείς θα προστατεύονται περισσότερο από ε, αναλυθείς πληροφορίες, από ψευδείς πληροφορίες ή από πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να, ανακαλύψουν από ποιον προέρχονται. Γιατί ε, ε, ε, τέτοιου είδους πληροφορίες τις βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Σετζήρη. Αντιλαμβανόμαστε πως το φαρμακευτικό πακέτο δεν θα περάσει μέσα στον 2009. Δηλαδή σίγουρα αν να γίνει κάτι θα γίνει επί Ισπανικής ε, Προεδρίας. Απλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσετε αυτό που έχω να σας πω, δηλαδή ότι πραγματικά υποβάλαμε αυτό το πακέτο μετά από πολύ προσεκτική εξέταση και χωρίς να θέλει να ανταποκριθεί ε, σε κάποια βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ορισμένων. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμα τομέα ο οποίος έχει καταλάβει και σε αυτή την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε ό,τι αφορά την νομοθεσία δηλαδή για τα χημικά και την ε, κατάσταση η οποία κυριαρχεί σε σχέση με αυτό το τομέα. Έχουμε να κάνουμε με τον κανονισμό REACH εδώ. Ε, η νομοθεσία λοιπόν για το REACH ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά δύσκολη, ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο ε, και ε, όποιος είχε συμμετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις πραγματεύσει, συγγνώμη, δεν μπορούσε να ξέρει ευθύ εξ αρχή πού θα κατέλεγαν αυτέ. Δηλαδή, όλοι τελικά οδηγηθήκαμε σε κάποιε εκπλήξει. Ε, το 2010 θα αποτελέσει ένα αποφασιστική σημασία έτος για την εφαρμογή του κανονισμού REACH. δηλαδή η αρμόδια αρχή για τα χημικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο νομοθέτης. Ε, και θα πρέπει να σας αναφερθώ σε ένα κάποιο ευτελές αλλά σημαντικό χρηματοδοτικό ζήτημα. Και να σας πω πώς τα έσοδα από τα τέλη τα οποία θα ε, θα εισπράττει εν λόγω αρχή αναμένονται ε, στα τέλη του 2010 και όχι στι αρχέ του έτου. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σημαντική χρηματοδότηση από την πλευρά τη ε, κοινότητα για το μεγαλύτερο μέρο του έτου 2010. Και κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα πρέπει να προβλεφθεί στον προπολογισμό. Δεν θα ήθελα τώρα να σας αποκρύψω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για, αυτή, για τα όσα προβλέπει ε, το Συμβούλιο, δηλαδή για μείωση του σχετικού προϋπολογισμού αυτής της υπηρεσίας κατά 5 ε, εκατομμύρια ευρώ. Ε, θεωρώ λοιπόν πως ε, αυτή η περικοπή των ε, κοντιλίων του προπολογισμού δεν είναι σωστή γιατί εμείς κατά τη σύνταξη του προπολογισμού αυτού κινηθήκαμε πραγματικά στο πλαίσιο των απολύτως απαραίτητων και καθόλου παραπάνω. Άρα λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω την εμφατική μου, την κατηγορηματική μου αντίθεση με αυτή την πρόθεση περικοπής από το του Συμβουλίου και θα ήθελα ε, Εσεί, από την πλευρά δηλαδή, τη Επιτροπή περιβάλλοντα, να συνταχθείτε με την Επιτροπή των Προπολογισμών ώστε να ε, μην ε, γίνει αυτό, να μην περάσει δηλαδή αυτό από την πλευρά του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να προβαίνουμε στην υιοθέτηση μια νομοθεσία και Κοινοβούλιο και Συμβούλιο η οποία θα θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηγετική θέση ε, σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τα χημικά, αλλά μετά όταν περνάμε στο επίπεδο της εφαρμογής ε, να, να, να, κρατάμε τα ε, κονδύλια κλειστά και να μην θέλουμε να προβούμε σε χρηματοδότηση. Όταν λέμε δηλαδή ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι και κάνουμε το πρώτο βήμα, τότε θα πρέπει να κάνουμε και το δεύτερο βήμα. Θα πρέπει να προβούμε και στην αντίστοιχη χρηματοδότηση. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το eco-design και την βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την μετάβαση σε μια ε, ε, οικονομία η οποία θα συνοδεύεται από λιγότερες εκπομπές τη του άνθρακα και ε, θα είναι πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την διαχείριση των πόρων θα πρέπει να αποτελέσει, σα το είπα και προηγουμένως, βασικό στοιχείο μιας μελλοντικής πολιτική για την οικονομία και στο πλαίσιο της Λισαβόνα. Και έχουμε λοιπόν εδώ ένα σχέδιο δράσης το οποίο ε, προβλέπει μια νέα βιώσιμη πολιτική για, το, για τα προϊόντα που θα οδηγήσει δηλαδή σε μεγαλύτερη ε, φιλικότητα προς το περιβάλλον των προϊόντων, ε, θα διασφαλίσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα των αντίστοιχων πολιτικών και ταυτόχρονα ένα σημαντικό τμήμα της βιομηχανικής πολιτικής από τη δική μας πλευρά ήταν η περαιτέρω προώθηση του eco-design. Ε, είχε επιτευχθεί ε, συνένεση σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ε, αυτό ήταν ένα θετικό μήνυμα, πράγμα που θεωρούμε πως θα μπορούσε να συνεχιστεί με περαιτέρω ε, προϋποθέσεις για ε, ε, ευρύτερες ομάδες προϊόντων σε ό,τι αφορά δηλαδή τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών. Επιτρέψτε μου όμως να πω πως εξεπλάγει λίγο με τη συζήτηση που έλαβε χώρα σε ορισμένες χώρες, ειδικότερα στη χώρα την οποία εγώ γνωρίζω καλύτερα, δηλαδή τη Γερμανία, σε ό,τι αφορά τους παλιάς τεχνολογίας λαπτήρα δεν ήξερα εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα πως αποτελεί αναπόστασμο τμήμα του πολιτισμού μας αυτός ο παλιάς τεχνολογίας λαπτήρα. Ε, δηλαδή από τη μία πλευρά μας λένε ότι αναγνωρίζουν τα όσα ε, συμβαίνουν θα πρέπει να αλλάξουν αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κινούμαστε τόσο αντιφατικά. Και θα υπάρξουν και άλλα πρόοδα τα οποία έχουμε συνηθίσει, τα οποία έχουν γίνει μέρος τη ζωή μα, αλλά τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα από ενεργειακή και περιβαλλοντική άποψη πιο αποτελεσματικά προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτού του είδου ε, ρομαντική, αν θέλετε, φλιάρια, ειδικότερα στη Γερμανία, ε, δεν, δεν μπορώ να την καταλάβω. Δηλαδή ε, ε, για κάποιου ε, αρθρογράφου, οι οποίοι από τη μία πλευρά αναφέρονται σε αυτούς τους παλιά τεχνολογίες λαμπτήρες και το πόσο ωραία και από την άλλη πλευρά μετά από ένα μήνα οι ίδιοι θα γράψουν ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε μια πιο οικολογική βιομηχανική πολιτική. Θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. εμεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχίσουμε την δική μας προσέγγιση. Και εάν όλα τα προϊόντα τα οποία, των οποίων η χρήση έχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μας διαχείριση ε, τεθούν στα αντίστοιχα ε, πρότυπα, δηλαδή ε, γίνουν όσο πιο ενεργειακά αποδοτικά γίνεται, τότε θα καταφέρουμε, θα έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο αντίκτυπο στους δικούς μας πόρους και ταυτόχρονα θα επιτύχουμε πως θα έχουν μικρότερο κόστος τέτοιου είδους ε, προϊόντα μέσω και μάκρο πρόθεσμα. Άρα λοιπόν δεν θα ήθελα να ε, να σας επηρεάσει όλη αυτή η συζήτηση, η ενόχληση που προκλήθηκε σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των ε, λαπτήρων τεχνιών παλαιάς τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το carbon leakage. Βρισκόμαστε εδώ ε, εν ώψη κάποιων πολύ σημαντικών αποφάσεων που θα ληφθούν ε, με βάση βέβαια και τα όσα θα συμφωνηθούν από τη δική σας πλευρά και στη Κοπενχάγη ούτω ώστε να μπορέσουμε τελικά να ε, κλείσουμε και αυτό το πακέτο σε ό,τι αφορά την διαρροή του άνθρακα, carbon leakage. Η διαδικασία επιτροπολογίας σκηνάει τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, άρα λοιπόν θα ενημερωθούμε αντίστοιχα και εσείς ε, προφανώς ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε ό,τι αφορά ε, τέτοιου είδους διαρροές και γι' αυτό κατά τη δική μας άποψη έως το τέλη του 2009 θα πρέπει να φτάσουμε σε οριστική λύση. Έχουμε μέχρι στιγμής εξετάσει 258 βιομηχανικούς τομείς και υποκλάδους. Αυτοί λοιπόν οι 258 τομείς ε, που αξιολογήθηκαν έχουν ε, καταδεικνύουν υψηλό ε, κίνδυνο σε ό,τι αφορά διαρροή άνθρακα και θα πρέπει κατά συνέπεια να τους διατεθούν και κάποια δικαιώματα εκπομπών ε, ατέλος. θα πρέπει τα ε, κάποια από αυτά τα τέλη να καταβληθούν παρόλα αυτά. Για παράδειγμα, ο τομέα τη παραγωγή ενέργεια δεν μπορεί να λάβει τέτοια ε, δικαιώματα ε, και άλλωστε έχουμε και κάποια benchmarks τα οποία εφαρμόζουμε, δηλαδή σχετικές μελέτε. Οπότε Ε, θεωρούμε πως θα κινηθούμε πολύ γρήγορα σε ό,τι αφορά την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μείωσης των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Έως λοιπόν το 2010 θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει και ε, εδώ τη συζήτηση, θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο εδώ την τεχνολογική ανάπτυξη και θεωρούμε πως θα οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ε, θεωρούμε πως το αντίστοιχο κόστος ε, μπορεί πράγματι να το αναλάβει η βιομηχανία μας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Τα θυμόσαστε ότι ε, σε πολλές και λύσεις που αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα. Ε, καταρχήν ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, έπεσε στην κρίση αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ο πρώτος κλάδος στον οποίο είδαμε να συμβαίνουν κάποια ανησυχητικά πράγματα. Αυτό ήδη είχε συμβεί το περσινό καλοκαίρι. Είδαμε να μειώνονται σε σημαντικό βαθμό οι πωλήσει εκεί. Ε, τελικά φτάσαμε σε μια αρκε... Ε, σχετική σταθεροποίηση, σταθεροποίηση συνόμιου του κλάδου μέσω και σχετικών ε, μέτρων για την ενίσχυση της υφιστάμενου στόλου μέσω για παράδειγμα απόσυσης παλαιών οχημάτων γιώταχη. Ε, αντιλαμβάνομαι πως πρόκειται για ένα κάπως αμφιλεγόμενο μέτρο είναι δύσκολο να επιτύχουμε μια ομαλή προσγείωση όταν θα ε, εκπνεύσουν και αυτά τα μέτρα. Αλλά είναι σημαντικό πως η αντικατάσταση παλαιών οχημάτων, δηλαδή παλαιότερων από 10 έτη με νέα οχήματα, ε, έχει και θετικό αντίκτυπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα όχημα το οποίο να κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον οποίο να μπορεί να συγκριθεί με ένα όχημα προ δεκαετίας ως προς την ε, αποδοτικότητά του σε σχέση με τα καύσιμα. Ε, δηλαδή σίγουρα υπάρχει εδώ ένα, μια θετική παράμετρο σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αυτοκινητοβιομηχανία, θα πρέπει να πούμε πως η νομοθεσία την οποία εμείς ε, αποφασίσαμε έχει δώσει εδώ την κατευθυντήρια γραμμή ότι δηλαδή η, η μείωση των εκπομπών του άνθρακα δεν μπορεί να καταστεί δυνατή, δεν είναι εφικτή με α, παραδοσιακές εντό εισαγωγικών τεχνολογίε, τεχνολογίες, ε, δηλαδή με κινητήρες καύσης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να προωθούμε την σταδιακή μετάβαση σε εναλλακτικέ τεχνολογίες ε, και κάτι τέτοιο είναι προφανώς σωστό, δεν έχουμε αντιρρήσεις να ενθαρρύνουμε δηλαδή την αυτοκινητοβιομηχανία να ακολουθήσει αυτή την οδό καθώς ε, μόνο ε, κάνοντας αυτό θα μπορέσει να είναι επιτυχής σε παγκόσμιο επίπεδο μακροπρόθεσμα. Όμως επιτρέψτε μου να πω να προσθέσω λοιπόν ότι και σήμερα μπορεί κανείς να αγοράσει ένα ε, αυτοκίνητο σχεδόν απαλλαγμένο από εκπομπές. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι εδώ στην αίθουσα οι οποίοι είναι αρκετά πλούσιοι για να αγοράσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ή μάλλον δεν έχουμε φτάσει. ο Όπου το φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκίνητο έχει μια τιμή η οποία να μπορεί να καταβληθεί από το μέσο πολίτη και από την άλλη πλευρά ε, ανταποκρίνεται και στις απαιτήσει ό,τι αφορά την κινητικότητα. Δηλαδή οι δυνατότητές του ε, απέχουν ακόμα πολύ από, τη, από τα όσα απαιτούμε, από τα όσα είναι αναγκαίο. Και η συγκέντρωση των ε, ε, προσπαθειών και της έρευνας ε, που γίνεται στην ε, μπαταρία και στη μεγαλύτερη δηλαδή αποδοτικότητα της μπαταρίας αυτών των οχημάτων θα, θα αποτελούσε πραγματικά μεγάλη έκπληξη το να μην επιτευχθούν πάρα πολύ μεγάλες πρόοδες σε αυτό το τομέα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αλλά δεν θα πρέπει, αυτό δηλαδή προσπαθώ να πω, να λέμε στους ανθρώπους ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Ότι δηλαδή το βράδυ θα βάζουν στην πρίζα το αυτοκινήτο και μετά θα μπορεί πάλι να α, τους μεταφέρει για μερικές εκατοντάδες ε, χιλιόμετρα. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα προβλήματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την απόδοση της ε, μπαταρίας, αλλά ε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, τα γνωρίζετε ίσως ο καταναλωτής απλώς τα γνωρίζει επαρκώς. Τελευταίο σημείο τώρα σε σχέση με αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που γίνεται στον ε, τομέα της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής και της, για το ζήτημα της General Motors. νομίζω πως και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τα όσα σας είπαμε με βάση αυτό το υπόβαθρο. Δηλαδή, η επιβλακτική στάση της General Motors στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε μια συμφωνία με τις ευρωπαϊκές χώρες ε, σχετίζεται και με το γεγονός αποτελεί στο πλαίσιο του δικού της ομίλου ε, εταιριών ε, την, τον κύριο παίκτη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Και είδαμε λοιπόν πως η πολιτική λοιπόν που ακολουθεί ε, στο Detroit General Motors ε, τους τελευταίους μήνους αποτελεί μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση από τα όσα έκανε μέχρι τώρα και κατευθύνεται περισσότερο προς την ε, ευρωπαϊκή στάση. Το σημειώνω απλά αυτό. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Το σημειώνω για να σας επιστήσω στην προσοχή ότι θα πρέπει να κρατάμε πάντα κατά νου τον ανταγωνισμό. Και θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μόνο εφόσον παραμείνουμε συνεπείς ε, στις ε, πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για αυτή την εξαιρετικά εκτεταμένη επισκόπηση που κάνετε στον κλάδο της βιομηχανίας και που μας θυμίζει αυτό που είπε πριν από λίγο ο Σουηδός Υπουργός για την ανάγκη να στραφούμε ε, προς μια οικο αποτελεσματική οικονομία. Θα σας δώσω το λόγο περιμένοντας την επιστροφή του Προέδρου της Επιτροπής μας. Θα σας παρακαλούσα να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας στο τρίλεπτο. Γιατί κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σε όλους να λάβουν το λόγο. Ξεκινάμε από την κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Είναι γεγονός ότι όλη αυτή η ανασκόπηση των διαφόρων φακέλων που, με τους οποίους ασχολείστε δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μην χάνουμε χρόνο. Θα είμαι σύντομη λοιπόν και θα μιλήσω μόνο για τα θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Μας είπατε ότι στην απομίμηση φαρμάκων δεν πήγαιναν άσχημα τα πράγματα στην καταπολέμηση του θέματος. Ξέρετε ότι είναι ένα επίγον ε, ζήτημα που ε, θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες. Πρόσφατα στη Γαλλία οι τελωνιακοί ε, κατάσχεσαν 13.000 ε, παραποιημένα φάρμακα. Ξέρετε ότι ε, η, καταπολέ... η παραγωγή της φαρμακοβιομηχανίας έγινε πολύ δύσκολη. Μέχρι να φτάσει από το, προϊόν, μέχρι να φτάσει στον ασθενή, περνάει από 30 ε, από 30 διαφορετικά χέρια. Άρα και ο έλεγχος της νόμιμης φαρμακοπαραγωγής δυσχεραίνεται. Πόσο μάλλον οι απομιμήσεις. Κύριε Επίτροπε, τώρα μπαίνω στην ερώτησή μου. Οι προτάσεις της Επιτροπής επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ακαιρεότητα του φαρμακείου, το packaging. Τι μπορούμε να κάνουμε η συναπόφαση παίρνει πολύ χρόνο. Πριν φτάσουμε σε μια οριστική απόφαση θα περάσει πολύ καιρό. Μπορείτε να εξετάσετε στο ενδεχόμενο αυτό κάποια ενδιάμεσα μέτρα. Δεύτερο, ε, το εμβόλιο κατά της ε, πανδημίας της γρήπης των χείρων. Ξεκινούμε να παίρνουμε τα στοιχεία από τους παρασκευαστές για το εμβόλιο αυτό. Χρειάζεται μια ε, επίγουσα διαδικασία. Εξετάζει η Επιτροπή την υιοθέτηση μια τέτοια ε, διαδικασία. Ε, Γνωρίζοντα ότι οι νέοι κανόνες στο Κοινοβούλιο του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχει θέματα επιτροπολογία. Ωστόσο, το δικαίωμα ελέγχου της επιτροπολογίας, δικαίωμα του Κοινοβουλίου που το θέλουμε και το κρατούμε, θα επιβαρύνει κατά ένα μήνα τουλάχιστον της προθεσμίας. Δεν μπορούμε όμω να χάσουμε χρόνο στο σημείο αυτό. Τι μπορείτε να μα προτείνετε, κύριε Πρόεδρε, ακριβώ για να υπάρξουν μέτρα που θα είναι μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά, θα μειώνουν το χρόνο και δεν θα ε, δυσχεραίνουν το δικαίωμα ελέγχου που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφόμου. Ε, κύριε Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον Επίτροπο και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πάντα εύκολο να συζητάμε με επιτρόπους όταν έρχονται στις συναντήσεις μας, αλλά αυτό που θέλω εγώ και που ενδιαφέρει και άλλα μέλη είναι πολλά και πραγματικά θα λυπηθούμε πολύ όταν σταματήσετε να ασχολείστε με τον τομέα αυτό. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, συνεχίσουμε, να συνεχίσετε να δουλεύετε στον τομέα αυτό όσο περισσότερο γίνεται. Στο πακέτο των φαρμακευτικών και σε άλλους τομείς, όπως αυτά που κάνετε για το πακέτο, για τα καλλιντικά, για την απαγόρευση ε, ε, τεστ ε, πειραμάτων σε ζώα λοιπά, Θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε κατά τη διάρκεια τη ε, θητεία σα. Καλύψατε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στην ομιλία σα. Εγώ θέλω να πω δύο-τρία πράγματα και κάποιε προτάσει ε, υγειονομική πολιτική που είναι ενώπιον του Κοινοβουλίου. Φαρμακοεπαγρύπνηση, φαρμακολογία, ενημέρωση των ε, ε, ασθενών. Η φαρμακοεπαγρύπνηση βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ε, μας έχει απασχολήσει πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων Βέβαια δεν προχωρήσαμε όσο θέλαμε, δεν πήγαμε παραπέρα. Ε, δεν είναι δικό σας λάθος, ε, είναι, δεν είναι δικό μας λάθος, είναι λάθος των κρατών μελών που δεν έχουν τα, σωστά μέσα για να προσφέρουν τα δεδομένα που χρειάζονται. Το μπαλάκι πήγαινε πέρα εδώ και στην πατρίδα μου ακόμα το ίδιο είναι, αλλά τι να κάνουμε, ε, πρέπει να σεβόμαστε μια σειρά υποχρεώσεων που έχει που έχουν τα πράγματα. Τώρα, η απομίμηση φαρμάκων. Στο παρελθόν είχαμε ετοιμάσει μια έκθεση που νομίζω ότι αποτελεί καλό κείμενο εργασίας. Το ανέφερε και η κυρία Γκροστέτ. Θέλουμε να προστατεύουμε τους ασθενείς και πρέπει να, και θέλουμε να εξασφαλίζουμε ότι η καταπολέμηση της, ε, των παραποιημένων φαρμάκων δεν ε, θα, θα συνεχίζεται, ιδίως ε, της των ασθενών ενδεχόμενος ε, το, το φαρμακευτικό προϊόν να μην δουλεύει σωστά ή να δημιουργεί ε, παρενέργειες. Πιο σύνθετο είναι το θέμα της ενημέρωσης των ε, ασθενών και πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος φωνάζει και αντιδρούν όταν ε, βλέπουν το θέμα της ενημέρωσης των ε, ασθενών και το ταυτίζουν με τη διαφήμιση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε, να ρυθμίσουμε εδώ θέματα ε, διαφήμισης. Υπάρχουν κανόνες που λένε ότι τα, τα φάρμακα δεν μπορούν, τα φάρμακα που δίνονται με συνταγή, τα συνταγογραφημένα φάρμακα δεν διαφημίζονται. Εμείς όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα. Υπάρχουν πληροφορίες σε μια σειρά περιοδικών, ε, ε, επιστημονικών περιοδικών, ε, άλλων περιοδικών και οι οργανώσεις ασθενών στην Ευρώπη τονίζουν ότι τα δικαιώματα των ασθενών πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα δικαιώματα, όπως και τα δικαιώματα του υγειονομικού προσωπικού. Πολλοί που ξέρουν αγγλικά και έχουν κομπιούτερ μπορούν να, στο, να βρουν τι πληροφορίε που χρειάζονται στην ιστοσελίδα στι ΗΠΑ. Πολιτείες. Ε, η Επιτροπή συζητά το ενδεχόμενο να, δει, να υπάρχουν πληροφορίε για ασθένειε, όχι για φάρμακα. Αλλά αν θε να βρει πληροφορίε για τι ασθένειε, πρέπει να ξέρει και τι φάρμακα αντιμετωπίζονται και πρέπει να έχει τι άδειε. Πιστεύω ότι έχουμε την υπηρεσία χορήγηση ε, αδειοδότηση φαρμάκου στο Λονδίνο. Στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη κατά βάση το θάψανε την πρόταση αυτή και αυτό είναι απαράδεκτο πιστεύω. Τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να περάσει αυτή η νομοθεσία είναι τα κράτη εκείνα που δεν θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση οι ασθενείς. Απαράδεκτο επαναλαμβάνω. Υπάρχει μια πρόταση που μπορεί να βελτιωθεί σίγουρα ε, αλλά γενικότερα θα ήθελα να τονίσουμε ότι είναι ντροπή που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για το θέμα της ε, ε, ενημέρωσης των ασθενών. Κάνουμε, μερικοί έχουν την εντύπωση ότι φροντίζουν περισσότερο τη, τα ζώα παρά τους ασθενείς. Άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες, σε δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά και σωματικά και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους δεν μπορούμε να παρα, να παραμερίζουμε τις προτάσεις αυτές. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από εσά να πείτε, να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη γιατί δεν κάνουν κάτι περισσότερο στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Ροτ και συμπαθάτε μας. Η κυρία Ρίστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να χαιρετήσω θερμά για την παρουσία του τον Επίτροπο Συμφωνώ και εγώ, χαιρετίζω και την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι συνάδελφοι. Βέβαια, όπω είπατε, δεν θα ολοκληρώσετε εσεί αυτή τη δέσμη μέτρων. Ευχαριστούμε και για αυτά τα οποία εξαγγείλατε. Ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνουμε ρεαλιστέ. Συμφωνούμε επί τη αρχή. Αλλά όταν έρχεται η ώρα τη προσγείωση και αλλαγή κάποιων νοοτροπιών, τα πράγματα είναι το πιο διστακτικά. Οπότε, για αυτή τη δέσμη τον για τα φάρμακα, πρέπει να μιστούμε γιατί ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η Φρανσουάζ Ροστέτ και η Ντάγμα Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει ευρύτερη συνέντευξη από το παρελθόν, από το 2003 στο Κοινοβούλιο. Είχαμε τότε περισσότερη απόκληση απόψεων, κάτι το οποίο δεν ωφέλησε ούτε τους ασθενείς, ούτε την βιομηχανία. Χρειάζεται καινοτομία πλευράς βιομηχανίας, αλλά χρειάζεται για τα γεννόσιμα φάρμακα επίσης ε, μια περισσότερη διείσδυση στην Ευρώπη. Όπως είπατε, χρειάζεται και διαφήμιση και ενημέρωση. Καμιά φορά αυτό το μιλήσετε σαν ταμπού και αυτό είναι κατανόητο, όπως είπε και η Ντάγμαρ. Μήπως γίνεται επίτροπε να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς μας και να προχωρήσουν προς ε, ένα πιστοποιημένο ε, website που να έχει την έγκριση των αρμοδίων οργανισμών. Να υπάρχουν οι πληροφορίες που χρειάζεται. Βέβαια, δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο ε, ίντερνετ, ε, ούτε 30% δεν διαβάζουν τις οδηγίες, αλλά ε, όσον αφορά δηλαδή τα, τα, τις άλλες πηγές πληροφόρησης, αλλά πάση τόσο όλο ένα για να ανεβαίνει η διείσδυση στο ίντερνετ, επομένω εκεί θα πρέπει κάτι να κάνουμε, ένα τέτοιο πιστοποιημένο website. Τώρα για τα παραγωγμένα φάρμακα, ε, είναι παλιό το πρόβλημα, τα είπε η κυρία Γκροστέτ, και εδώ το συζητούμε συνέχεια. Έχουμε κατασχέσεις, όλα ένα και περισσότερες τέτοιων φαρμάκων, ε, τριπλάσεις από ό,τι στο παρελθόν. Είναι μάστιγα αυτά τα φάρμακα. Οπότε για πέστε μας πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο συντοπιμένους πιο ευαίσθητους τους πολίτες όσον αφορά την, την πληροφόρηση που πρέπει να έχουν, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να ξέρουν τι κινδύνους ενέχουν αυτά τα φάρμακα. Ξέρω ότι έχει χτενιστεί ή παραχτενιστεί το κείμενο το αρχικό της Κομισιόν, οπότε όπως τον η Ντάγμαρ πέστε μας τι θα κάνουμε με αυτή τη δύσκολη μάχη, τον πόλεμο κατά των παραπημένων φαρμάκων. Πώς θα συνεργαστείτε με το Συμβούλιο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και όσον αφορά τα καλλιντικά. Είναι εγκάρσιο αυτό το θέμα, αφορά όλα τα χαρτοφυλάκια στην Επιτροπή. Ε, τώρα μίλησε περισσότερο, αλλά πριν μίλησε λιγότερο από ό,τι δικαιούμε. Να δούμε επίσης τι θα γίνει με τις παράλληλες εισαγωγές. και βέβαια ταυτόχρονα με τον πόλεμο κατά τι παραπείσει να είμαστε και αποτελεσματικοί στην πολιτική μα. Ευχαριστούμε κύριε Ρίση και τώρα έχει το λόγο ο κύριο Σλίτερ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φερχόγγεν για την ε, παρουσίαση που έκανε. Όταν μιλάμε για την βιομηχανία στην Ευρώπη είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες. Μήπως θα μπορούσε. Μήπως θα μπορούσε να μιλήσει ε, περισσότερο για τα θέματα της αποτελεσματικότητας και της επίδοσης των ε, κινητήρων στα οχήματα. Χαίρο που μιλήσατε για την εξοικονόμηση που μπορούσαμε να πετύχουμε στην χημική βιομηχανία ε, και την ανάγκη να, να λειτουργήσει πραγματικά το REACH. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε το, τον προπολογισμό εκεί. Για να υλοποιηθεί σωστά το ΡΙΤΣ χρειάζονται περισσότερα χρήματα και πρέπει το Κοινοβούλιο να το συμφωνήσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θέλω να πω και κάτι άλλο για την φαρμακοβιομηχανία. Δεν κατάλαβα πρέπει να σας πω αυτό που είπατε. Μιλήσατε, είπατε ότι δεν θέλετε διαφήμιση, αλλά μετά μιλήσατε για γκρίζες ζώνες. Κάποια στιγμή είπατε ότι υπάρχουν κάποια φυλάδια που απευθύνονται σε ιατρούς, σε κάποια περιοδικά ε, μπορούμε να δούμε αναφο... σχετικές αναφορές. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι ένα γερμανικό γυναικείο περιοδικό από τη φίλη μου τη Γερμανίδα το πήρα που έχει μια πάντα, αυτό το περιοδικό, ένα πάντα ένα τμήμα ε, υγεία. Και εδώ έχει διαφήμιση στον τομέα υγεία. Πώς μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Μιλήσατε για γκρίζε ζώνες. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν τηρούν ορισμένες διατάξεις. Μήπως θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε ό,τι αφορά αυτές τις γκρίζε ζώνες, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο θέμα για τα παραποιημένα φάρμακα. Πραγματικά είναι φοβερό να, μπορεί να, να ξέρει ότι μπορεί να βρει οπουδήποτε οτιδήποτε. Δεν ξέρει αν η δόση που περιέχει το συγκεκριμένο φάρμακο είναι η σωστή, αν πρέπει να το καταπιείς ή να το μασεί Υπάρχουν ε, μια σειρά προβλημάτων με τα φάρμακα αυτά. Μπορεί να έχουμε ε, πολλές κατασχέσεις, ε, τον περασμένο μήνα είχαν κατασκευή στην Ολλανδία φάρμακα από την Ινδία και την Βραζιλία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ε, βρούμε μια ισορροπία ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να μας δημιουργήσουν τρομερούς φόβους. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύρια Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να μιλήσω για το φαρμακευτικό πακέτο. Ιδίω για την οδηγία για τα παραποιημένα φάρμακα. Άκουσα προσεκτικά τα θέματα που αναφέρατε και τα λόγια σας Καταλαβαίνω τη θέση σας πρέπει να σας πω, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ταυτόχρονα ότι ζούμε σε άλλες εποχές. Ο χρόνος που έχει το Κοινοβούλιο είναι χρόνος τον οποίο πρέπει να σκεφτούμε και τα, θύμητα, τα θύματα. Στην περίπτωσή μας τα θύματα των παραποιημένων φαρμάκων. Συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να υπάρχει μια δράση σε προληπτικό επίπεδο. Ναι, αλλά το Κοινοβούλιο, το, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κάνουν, ε, έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι θα πρέπει να αλλάξετε κάπως την πρότασή σας ενώπιον του Κοινοβουλίου, γιατί την αλλάξατε ήδη και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του Κοινοβούλου για να κάνει τη δουλειά που κάνει, που είναι αρμόδιο να κάνει. Να κάνω κάποια άλλα σχόλια τώρα. Μας προτείνεται μια οδηγία σημαντική σαν Επιτροπή. Αυτό το, το αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό το κείμενο. Σήμερα ένας ασθενής, ο οποίος δεν έχει καμία εγγύηση όταν ε, ότι αγοράζει ένα αυθεντικό φάρμακο όταν πηγαίνει σε ένα φαρμακείο. Δεν θέλουμε να χάσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στην ε, λειτουργία των φαρμάκων. Άρα θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια. Αυτό προτείνει η Επιτροπή να γίνει με μια σειρά μέσων. Εντοπισμός των ε, πυλών εισόδου των πλαστών φαρμάκων, ε, παρεμπόδιση της τροφοδότησης, ρυθμιστική πολιτική που εξασφαλίζει την καταχώρηση κάθε βήματος και επιτρέπει έτσι να εντοπίζεται ένα παραποιημένο φάρμακο από την παραγωγή μέχρι την τελική αγορά του από τον ε, ε, ασθενή. Εγώ υποστηρίζω τις προτάσεις της Επιτροπής και πιστεύω ότι είναι θέματα που θα έπρεπε να τα σκεφτούμε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο, επαναλαμβάνω. Δεδομένου ότι δεν έχω πολύ χρόνο, θα αφήσω τα παραδείγματα που ε, θα έπρεπε να σας σχολιάσω μέσα και τα οποία θα αναφέρονται σε συγκεκριμένες τοπολογίες. Από τον ορισμό, τι είναι παραποιημένο φάρμακο, κάτι πολύ σημαντικό, διότι μόνο ένα σαφής ορισμός θα μπορέσει να οδηγήσει στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων κατά της, ε, του αδικήματος αυτού. Και τούτο μόνο εάν υπάρξει καλύτερη διεθνής συνεργασία θα επιτευχθεί. Έχουμε δύο δυνατότητες. Είτε ε, δεχόμαστε την τον υφιστάμενο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή πηγαίνουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εξετάζουμε τον ευρωπαϊκό ορισμό. Μιλάμε μόνο για τις ενεργές φαρμακευτικές ουσίες ή πρέπει να ε, περάσουμε και άλλες ε, έννοιες μέσα στον όρο του φαρμάκου αυτού. Δεν έχω άλλο χρόνο βλέπω και τελειώνω λέγοντας υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Φερρυπίν, πώληση μέσω ίντερνετ. Κλείνω. Θα ήθελα να σας πω κύριε Αντιπρόεδρε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο ταχύτερη και καλύτερη δουλειά γίνεται στην οδηγία αυτή με τους κοιόδους εισηγητές για να βελτιώσουμε την πρόταση που μας έχετε υποβάλει προς όφελος των ασθενών και των πολιτών γενικότερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα παραποίησης φαρμάκων στην αγορά. Ο κόσμος υποφέρει, είναι θύματα και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά βάση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιαννάκου. Για κουδάκι, Συγγνώμη, κυρία Γιανακουδάκη. Sorry, um, I'm going to be passing my question on to my colleague. Ο, συνάδελ, ε, ο συνάδελφος ε, θα θέσει το ερώτημα. Περνάω την ερώτηση στον συνάδελφο. Γιατί έχει ήδη και κάποια κύριος Κάλαναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα ρωτήσω κάτι σχέση με τα όσα στην αρχή μας είπατε, Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω που ήρθατε και μας τα είπατε τόσο ξεκάθαρα όπως πάντα κάνετε. Δεν, δεν αλλάξατε την στάση και συμπεριφορά σας ούτε σήμερα. Είπατε για τους λαμπτήρες, είπατε για αυτές τις ρομαντικές φλαγίες που έχουν προηγηθεί, είπατε για αυτή την ιστερία που αφορά αυτή την υπόθεση. Βέβαια, με πολλά πράγματα ευσταθούν εδώ πέρα, δηλαδή θέλουμε όσο γίνεται συντομότερα να πάμε σε πιο αποδοτικές, ε, αποδοτικές λάμπες. Όμως προσοχή, μην, μην, μην ε, βιαζόμαστε γιατί έτσι οι πολλοί καταναλωτές γίνονται δύσπιστοι όσον αφορά τις προτινόμενες εναλλακτικές γιατί πολλές φορές ε, οι καινούργιες λιχνίες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο οι κλασικές η ένταση του φωτός δεν βοηθάει ε, να δουλέψει κανείς ή να μπορεί να χαμηλώσει τα φώτα με, με, με διακόπτες. Λοιπόν, ελπίζω όλα αυτά να τα λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν πριν απαγορεύσει τελείως τους, ε, τις κλασικές λάμπες και ο κόσμος ε, πάει να αγοράζει μαζικά για να ε, τους κρατήσει, ούτω ώστε να το χρησιμοποιεί μια που οι καινούργιοι λαμπτήρε δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικοί όσο οι παλιοί. Τώρα για τα αυτοκίνητα, αυτά που μα είπατε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και στέκομαι στο εξή. Είπατε ότι ακόμα δεν φάσαμε στην φάση που η τιμή των περιβαλλοντικά φιλικών αυτοκινήτων είναι λογική. Εξαρτάται από τον ορισμό που δίνει κανεί ε, στο, στο, στο πράσινο, στο οικολογικό αυτοκίνητο. Τι λέτε για την μείωση εκπομπών όσον αφορά τα ελαφρά φορτηγά, τα ημιφορτηγά, αυτά τα βαν και τα μίνι μπας. Για πέστε μας, πότε το Κοινοβούλιο θα λάβει το κείμενο της σχετικής πρότασης Κομισιόν. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Και τώρα, η κυρία Ρόσμπαχ θα υποβάλει την τελευταία ερώτηση για αυτόν τον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Επανειλημμένα, τα έχουμε αναφέρει. Δεν, δεν έκλεισε το μικρόφωνο τώρα η Μιλήτρια. Αναφέρατε προηγουμένως το θέμα αυτών των φαρμάκων που ε, προέρχονται από την από Ανατολία. Τι θα γίνει με τα φάρμακα αυτά, τι θα γίνεται με τα φάρμακα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό. Για πέστε Για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Μιλούμε για μέτρα απαγορευτικά ε, όσον αφορά τις λιχνίες. Έχουμε τώρα τέσσερα διαφορετικά χρώματα ε, για αυτές τις νέες οικονομικές λάμπες, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παντού. Δεν είναι αρκετό το φως που δίνουν. Μήπως γίνεται να δούμε καλύτερα πιο φιλόδοξα αυτά τα μέτρα. Απαντήστε κύριε Πίτρο, αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την τα ερωτήματα τα οποία ε, αναφέρθηκαν ε, στα φαρμακευτικά και ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της, των παραβημένων προϊόντων στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χωστέ και άλλοι αυτό, τα όσα προβλέπουμε νομοθεσία μπορεί να αναφέρεται μόνο προφανώς σε νόμιμα στεβάσματα. Δεν μπορούμε να έχουμε διατάξεις για παράνομα στεβάσματα, ε, καθώς αυτά απαγορεύονται ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την ε, νομοθετική πρόταση είναι ότι στην νόμιμη αλυσίδα προώθηση ε, πώληση δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανακύπτουν παράνομα στεβάσματα όπου και αν αυτά έχουν παρασκευαστεί. Ε, και ε, θέλουμε με αυτή την πρόταση να αξιοποιήσουμε στο ακέραιο όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε, ώστε να μπορούμε να επαληθεύουμε την ακαιρεότητα και ε, την, ε, το ότι δεν έχει υποστεί κανένα είδου φθορέ ή ε, συσκευασία κάποιου συσκευάσματο. Άρα λοιπόν με τα όσα προβλέπουμε διασφαλίζουμε δύο πρόγραμματα. Πρώτον το σκευάσμα, το προϊόν το οποίο λαμβάνει ο καταναλωτή στο τέλο είναι σίγουρα 100% το προϊόν το οποίο επιθυμεί, αυτό δηλαδή το οποίο ζήτησε να λάβει και το δεύτερο ότι η συσκευασία δεν υπέστη φθορέ από την μετάβαση δηλαδή στον πολιτή προ τον ε, καταναλωτή. Δηλαδή δεν ανοίχθηκε ποτέ. Και αυτό ε, είναι σημαντικό γιατί όπω ήδη είπε η κυρία Ρή ε, στην νόμιμη πώληση των ε, φαρμακευτικών συμβαστημάτων έχουμε πραγματικά πάρα πολλά στάδια στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ε, και εγώ είχα εκπλαγεί ο ίδιος όταν ε, ενημερώθηκα σχετικά. Πράγματι, ενδεχομένως από οικονομική άποψη είναι ενδεχομένως αμφιλεγόμενη με τέτοια πολιτική, αλλά αυτή ισχύει εντάξει, μπορούμε να αναλογιστούμε το πώς ε, μπορούμε να λάβουμε άλλα μέτρα και είμαι ανοιχτό σε προτάσει, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχουν και από τεχνική άποψη άλλες δυνατότητες ούτως ώστε να μπορέσουμε να ε, διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα αυτό, δηλαδή ότι δεν έχει υποστεί η συσκευασία, πέρα από τα όσα προβλέπουμε ήδη και την επαλήθευση της αυθεντικότητας. Ε, δηλαδή, έτσι όπως θα ισχύει το σύστημα, ε, το κουτί το οποίο δίνεται σε εσά, ε, δηλαδή με ένα στέβασμα ε, από το φαρμακείο, αυτό θα πρέπει κατευθείαν να σαρωθεί από ένα μηχάνημα το οποίο ακριβώς θα ενημερώνει και θα διασφαλίζει ότι τότε από τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής έφυγε την τάδε ημερομηνία του εν λόγω στέβασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε από εκεί και μετά προφανώς ο ορισμός της παραποίησης ε, προφανώς και αναφέρεται στις δραστικές ενεργές ουσίες. Ε, όταν έχουμε να κάνουμε με φάρμακα, έχουμε να κάνουμε κυρίως προφανώς με τις δραστικές ουσίες οι οποίες ε, την χάνουν εδώ παραποίησης, γιατί αυτές είναι που κοστίζουν και τα χρήματα. Τώρα, εδώ υπήρχε και το ενδιαφέρον ερώτημα, κυρία Ρωσά, προς το τέλος δηλαδή των παρεμβάσεων, που μας ε, πηγαίνει πολύ πιο μακριά από το βασικό ερώτημα. Δηλαδή, σχετίζεται με, τη μεταχείριση παραδοσιακής, ε, παραδοσιακών συσκευασμάτων, ιατρικών σκευασμάτων ή σκευασμάτων από άλλη ε, μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, και από άλλες χώρες του κόσμου όπως ε, συμβάσματα από την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία. Ε, αυτό θα πρέπει να μας αποσχολήσει γιατί κανονικά δεν είναι συνταγογραφούμενα τα εν φάρμακα. Και στον ελόγο κανονισμό τέτοιου είδου φάρμακα καλύπτουμε. Δηλαδή μόνο συνταγογραφούμενα. Δεν κάνουμε λόγο για τα μη συνταγογραφούμενα. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα παραδοσιακά φάρμακα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι πάντοτε τόσο ακίνδυνα όπως μας ενημερώνουν κάποιες φορές οι παρασκευαστές τους. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ινδικά φάρμακα, της δηλαδή τη παραδοσιακής ειδική ιατρικής, ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, σαφώς επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες ε, μάλιστα εμφανίζονται σε συμπυκνωμένη μόρφη ε, και που υπερβαίνουν τις ανοχές του οργανισμού ε, πολλές φορές. Και παρόλα αυτά κυκλοφορούν εδώ και 50 χρόνια στις αγορές μας χωρίς να έχουν οδηγήσει σε πραγματική, σε, πραγματικές καταστροφές, δηλαδή σε πραγματικές συνέπειες. Άρα λοιπόν ε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε να κάνουμε ακριβώς με παραποίηση, αλλά με το ζήτημα του τελικά του τι θα επιτρέπεται και τι όχι να κυκλοφορεί στις αγορές μας. Ε, σε ό,τι αφορά την παραποίηση, ε, δηλαδή για τις εισόδου, οδού, αυτή μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των διοκτικών αρχών, των τηλεωνιακών αρχών και των αρχών παρακολούθησης της αγοράς και βέβαια το βασικό πρόβλημα παραμένει στον τομέα των παραποιημένων φαρμάκων ότι σε κάποια μέρη του κόσμου παρασκευάζονται παράνομα φάρμακα τα οποία προορίζονται για τις στοχόρτες χώρες ε, του κόσμου αλλά τελικά ε, βρίσκουν τον δρόμο τους και καταφέρουν να διεισδύσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή βέβαια κάποια από αυτά ένα μέρος τους παρασκευάζεται και στην ίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ένα μεγάλο μέρος αυτών ε, των ε, συμβασμάτων που παρασκευάζουν δηλαδή παράνομα προορίζονται για φτωχέ χώρε, για παράδειγμα για την Αφρική. Αλλά τελικά καταλήγουν και στην Ευρώπη, όπου το απαντούμε. Αλλά δεν προορίζονταν για την Ευρώπη. Ε, ε, φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία παρασκευάζονται παράνομα με στόχο για προώθηση δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο λίγα τα οποία είναι ιδιαίτερα ακριβά και τα οποία θεωρούνται ε, φάρμακα lifestyle ας το πούμε έτσι ε, και κάτι τέτοιο αντιλαμβανόμαστε το γιατί παρασκευάζονται τέτοιου είδου φάρμακα. Δηλαδή, αν, όταν υπάρχουν δηλαδή ε, φάρμακα των ε, αξίας 120 ευρώ ανασυσκευασία τα οποία απολούνται ε, παραβημένα για 8 ευρώ σε μια φτωχή αφρικανική χώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούμε, εγκρίνουμε κάτι τέτοιο, το κάθε άλλο. Πάντως, Ε, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε συγκεκριμένα συμβάσματα σε συγκεκριμένε περιοχέ. Δεν είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε ό,τι αφορά τι αρχέ αδειοδότηση και τι αρχέ παρακολούθηση τη αγορά. Ε, να του επιτρέψουμε να δραστηριοποιηθούν περισσότερο εκεί που πρέπει. Καθώ ειδικότερα οι φτωχότερε χώρε δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ακολουθήσουν τις διαδικασίες τις οποίες προβλέπουμε εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν όμω υπάρχουν δικέ σα προτάσει για να βελτιώσουμε τα όσα ήδη προτείνουμε, παρακαλώ, δηλαδή είμαστε πολύ ανοιχτοί. Σε ό,τι αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση είμαστε σύμφωνοι. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών, σα ευχαριστώ ε, για τις ε, παρατηρήσεις που κάνατε εδώ, η κυρία Ροτ Μπέρεντ και άλλοι συνάδελφοι, ε, η μόνη παράκληση από την πλευρά μου είναι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με την δέουσα αντικειμενικότητα και να μην υποβαθμίσουμε ε, τα όσα αφορούν τη βιομηχανία. Γιατί τα πράγματα είναι όπως τα περιέγραψε η κυρία Ρόντ Μπέρεντ. Οι άνθρωποι έχουν την πρόσβαση στις ε, πληροφορίες, αλλά είναι τέτοιου είδους οι πληροφορίες ε, έτσι ώστε να μπορούν να ξεχωρίσουν αν πρόκειται για πραγματική ενημέρωση ή διαφήμιση. Δηλαδή τα όσα βλέπουμε στο ίντερνετ από τους α, Αμερικανούς ε, ε, παραγωγούς από την Αμερικανική φαρμακομηχανία βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα, ε, στις προποθέσεις που έχουμε θέσει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δηλαδή στις ε, ΗΠΑ δεν έχει απαγορευτεί η διαφήμιση. Άρα λοιπόν έχει κανείς πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Και ο καθένας που έχει έναν υπολογιστή έχει πρόσβαση. Αλλά άμα ε, λέμε ότι σε 20 χρόνια θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούν να, να διαχειριστούν, ε, για παράδειγμα, τα νέα μέσα τεχνολογίας, τότε απαντάστε, προφανώς και θα μπορούν να το κάνουν. Άρα λοιπόν δεν είναι το ζήτημα εδώ ε, να ασχοληθούμε με, με αυτό το τομέα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, έχουμε να κάνουμε και με ζήτημα δημοσιογραφικής ηθικής. Πολύ σαφώς. Δηλαδή, αν ε, μιλήσουμε με εκδότες από εφημερίδες, από περιοδικά και ούτω καθεξής, γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα δύναμα σημεία των εντύπων τους. Αυτά που αφορούν την υγεία, τα, τα οχήματα και τον τουρισμό. Γιατί, Γιατί ο εκδότης δεν γνωρίζει ποτέ με βεβαιότητα κατά πόσο τα άρθρα τα οποία έχουν επηρεαστεί, δηλαδή από συγκεκριμένα επαγγελματικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να το διαπιστώσει εύκολα κανείς. Εδώ στην Επιτροπή σας, δεν θυμάμαι αν ήταν κάποια άλλη, όταν είχαμε συζητήσει το ζήτημα της ενημέρωσης των ασθενών, την ίδια ημέρα στη μεγαλύτερη ε, γερμανική εφημερίδα 5 εκατομμύρια ε, είχα μια ολόκληρη σελίδα από έναν καθηγητή ιατρικής ο οποίος τασόταν υπέρ της χρήσης ενός συμβολίου κατηγορηματικά μάλιστα για την ε, ε, για την καταπολέμηση του Καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και δεν αντιλαμβανόταν δηλαδή κανείς, δεν αναφερόταν μάλλον ε, πουθενά ότι ε, αυτός ο επιστήμονας εργαζόταν για την ελογοφαρμακομηχανία παρότι ήταν σαφές από το περιεχόμενο. Άρα λοιπόν τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ε, εδώ μια ρύθμιση η οποία θα καλύπτει και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή όχι μόνο της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και του εκδοτικού τομέα, του εκδοτικού κλάδου ε, για να μπορούμε να επιτύχουμε μια σωστή ρύθμιση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να φτάσουμε σε καμία άλλη ρύθμιση εκτός από αυτή του να έχουμε μια σχεδόν απόλυτη λογοκρισία και έναν απόλυτο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης σε αυτό το τομέα. Ε, αυτός μόνο, αυτή μόνο εναλλακτική υπάρχει για να ε, οδηγήσουμε στο να, στο να ε, καταστραφεί τελικά αυτή η γκρίζα ζώνη της ενημέρωσης. Αν η φαρμακομηχανία αρχίσει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα, δηλαδή δεν καταστατική τις σχετικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών, τότε θα πρέπει να μας προτείνει μια σαφή ελέγξιμη και διαφανή οδό. Ένα σαφή δηλαδή και διαφανή τρόπο. Και αν υπάρχει ένα τέτοιο τρόπο, σα έρθει να μας τον προτείνει. Ε, τώρα, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό που υπόθηκε στο συγγνώμη, ένα συνάδελφο δεν θυμάμαι ποιο πρότεινε κάτι για μία ιστοσελίδα. Κυρία Ρή. Ναι. Ε, θεωρώ πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και ε, σας καλώ και εσάς να τη σκεφτείτε. Μπορούμε να την ε, υλοποιήσουμε συμπληρωματικά. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε δηλαδή δυνατότητες ενημέρωσης ουδέτερες, στις οποίες δηλαδή δεν εμπλέκονται κανένας είδους επαγγελματικά συμφέροντα. Δηλαδή ούτε συμφέροντα εκδοτών, ούτε συμφέροντα φαρμακοβιομηχανιών ή πολιτών φαρμακευτικών ε, να υπάρχει δηλαδή μια ουδέτερη αρχή η οποία θα διαθέτει κάποιες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες ελεύθερες για το ευρύ Ε, θεωρώ πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση αυτή ως ε, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε συμπληρωματικά. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω κάτι στην κυρία Κλωστέτ σε ό,τι αφορά το ζήτημα με τα εμβόλια. Ε, προφανώς υπήρξε στο παρελθόν μια διαδικασία εδώ η οποία δεν ήταν ικανοποιητική 100%. Θεωρώ πως μπορούμε και θα πρέπει να βρούμε μια λύση εδώ η οποία θα διασφαλίσει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να μπορεί να παρεμβαίνει ε, ε, για την περίπτωση, ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι η υιοθέτηση νομοθεσίας για τα εμβόλια να μην ε, προσκρούει σε εμπόδια σε ό,τι αφορά την ταχεία δηλαδή οθέτηση. Επιτρέψτε μου να πω πάντως κάτι σε σχέση με την εμπειρία που έχω σε αυτό το τομέα. Εγώ ως πολιτικός ο οποίος δεν έχει σπουδάσει φαρμακολογία δεν μπορώ να εναντιωθώ στις συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Δηλαδή, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Μιλάμε δηλαδή για την έγκριση ενός ε, συνταγογραφούμενου φάρμακου, ε, το οποίο ε, κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στις αγορές μας. Κάποιοι λένε λοιπόν τώρα ότι είναι ασφαλές αυτό, κάποιοι ότι δεν είναι. Εγώ ως πολιτικός πώς μπορώ από ηθικής άποψης δηλαδή να αναλάβω την πρωτοβουλία και να πω ο Τάδε ή ο Δίνα έχει δίκιο. Δεν μπορώ εγώ ποτέ να κινηθώ ενάντια στη συμβουλή, στη, γνωμοδότηση τη, της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να ε, εγκριθεί αυτό το φάρμακο, θα το γίνει. Αν πει όχι, δεν θα εγκριθεί. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν βλέπω καμιά άλλη λύση για μένα να, να εναντιωθώ ε, στην γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής αυτής. Ε, δεν μπορώ να αναλάβω το ρόλο ενός φαρμακολόγου και να αρχίζω εγώ να συντάσσω τέτοιου είδους εκθέσεις, τέτοιου είδους μελέτες. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη δυνατότητα για μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη της Εμιστημονικής Επιτροπής. βρείτε μου έναν τρόπο ε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά, για παράδειγμα, σε περίπτωση σε ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει, τι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή για να λύσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτως ώστε να δεσφαλίζεται και σε πολιτικό επίπεδο ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να παρέμβει. Α, και ο κύριος νομίζω. Αυτό με το λαπτήρες. Εντάξει, ε, δεν μπορούμε να το επιτύχουμε μέσα σε μια μέρα. Και ε, ούτε άλλωστε αποφασίστηκε έτσι εδώ και χρόνια έχει δοθεί δημοσιότητα και υπήρξε, υπήρξαν συνενέσεις και σύμφωνες απόψεις υψηλού επίπεδου και ευρέως δημοσιευμένες. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν τώρα ε, γιατί έχει κινητοποιηθεί ε, μια τέτοια αντίθεση, αλλά πραγματικά κάτι τέτοιο με κάνει πολύ επιφυλακτικό. Πάντως εγώ επαναλαμβάνω, θα πρέπει να κάνουμε επιτέλους ένα αποφασιστικό μεγάλο βήμα κατά την καταστροφή του πλανήτη μας, ε, κατά των κλιματικών μεταβολών. Δεν μπορούμε όμως να ισχυριζόμαστε όλα αυτά και από την άλλη πλευρά να λέμε ότι δεν θα πράξουμε τα όσα είναι απαραίτητα. Όχι, ως πολιτικοί θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ε, προβούμε σε αυτά που πρέπει να προβούμε και να λάβουμε αυτή τη στάση απέναντι στους ε, πολίτες μας. Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο δεν αναφέρθηκα σε φιλοπεριβαλλοντικά αυτοκίνητα, αναφέρθηκα σε αυτοκίνητο χωρί εκπομπέ με σχεδόν χωρί εκπομπέ. Υπάρχουν κάποια περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικά αυτοκίνητα που μπορεί κανεί να υπολογίσει κατά πόσο είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά. Αλλά ένα αυτοκίνητο χωρί εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, σχεδόν χωρί εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, είναι ήδη από τεχνητή άποψη εφικτό, αλλά δεν ε, ε, ε, έχει επαρκώ χαμηλή τιμή. Άρα λοιπόν εγώ προβλέπω ότι στο μέλλον θα έχουμε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα με υβριδικό κινητήρα και πιστεύω πως οι πόλεις θα αρχίσουν να κινούνται καταρχήν προς τη λύση της ε, υποχρεωτικής ε, χρήσης ε, οχημάτων με ηλεκτροκινητήρα μέσα στην, στο κέντρο της πόλης και από εκεί μετά όταν μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουν αυξηθεί και αντίστοιχα οι αποθηκευτικές δυνατότητες δηλαδή ε, για τα χιλιόμετρα των ε, σχετικών αυτοκινήτων να ε, καταστεί περισσότερο πραγματικότητα το αυτοκίνητο αυτού του είδους με βέβαια με αντίστοιχες ανάγκες περισσότερης τροφοδοσίας με ρεύμα, με ηλεκτρική ενέργεια το οποίο έχει παραχθεί και αυτό με φιλεφορικό τρόπο. Τώρα σε σχέση με περισσότερες προτάσεις δεν έχουμε λάβει ε, κάποια πρόταση ούτε έχουμε ετοιμάσει ε, προτάσεις σε ό,τι αφορά δηλαδή τα βαν και τα μίνι, πούλμα μίνι λεωφορεία. Ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, ε, την κατεύθυνση δηλαδή του στόχου της επίτευξης μείωσης των εκπομπών όλων των ειδών των οχημάτων, κάτι δηλαδή που ισχύει αυτονόητα και ε, ελαφρά φορτηγά, βάνς ε, και ούτω καθεξής. Απλά το ζητούμενο εδώ είναι το να δούμε ε, ποια είναι σωστή χρονική συντηρία και το ποιο ποιος ενδιάμεσος χρόνος θα πρέπει να δοθεί στη μηχανή. Θεωρώ πως δεν είναι ευνοϊκή αυτή τη στιγμή η συντηρία γιατί οι αυτοκινητομηχανίε, οι οποίε αυτή τη στιγμή έχουν ε, πολύ λίγα κονδύλια στη διάθεσή του σε σύγκριση με άλλε περιόδου, δεν θα ήταν σε θέση καν να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο. Θα δούμε ε, θα συνεχίσουμε να προσέχουμε αυτό το ζήτημα, αλλά προφανώ και συντάσσω μαζί σα ότι θα πρέπει να προωθηθεί εδώ αυτό ο στόχο ε, τη ε, μείωση των κομπών διοξιδίου του άνθρακα όλων των ειδών μεταφορά, δηλαδή οδικών, σιδηροδρομικών, αέριων, πλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή. Έχουμε μισή ώρα, 35 λεπτά στη διάθεσή μα, κύριε συναδελφοί. Θα δώσω το λόγο σε όσο περισσότερους από εσά γίνεται, αλλά θα σας παρακαλούσα να μιλήσετε μόνο 1,5 λεπτό ο καθένας για να μπορέσουμε να κλείσουμε. Γιατί είσαστε πολλοί που θέλετε το λόγο. Ο κύριος Φίλνερ, καταρχάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγητής και είναι δύσκολο να μιλήσω σε 1,5 λεπτό. Τέλος πάντων, χαίρο που ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε στην Επιτροπή και χαίρο που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόταση, το ταχύ, να υπάρξουν προτάσεις το ταχύτερο δυνατόν για το θέμα της ενημέρωσης των ε, ασθενών και για να ενισχύσουμε τη γνώση του ασθενή. Ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο, αυτό είναι γνωστό για όλου. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι απαράδεκτο να μην έχουν στη διάθεσή του τι πληροφορίε αυτέ οι ασθενεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό περιμένουμε ε, σχετικές προτάσεις, 8 χρόνια από ό,τι θυμάμαι και δεν νομίζω ότι μόνο εμεί περιμένουμε. Ε, το περιμένουν οι ασθενεί, οι οργανώσει των ασθενών, Κανείς δεν είναι ικανοποιημένο από την υφιστάμενη κατάσταση. Βέβαια, από χώρα σε χώρα το σύστημα είναι διαφορετικό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο ασθενή δεν έχει ενημέρωση στις πληροφορίες, αν δεν έχει ίντερνετ, αν δεν ξέρει καλά αγγλικά. Ε, καταλαβαίνουμε ότι οι προτάσεις αυτές ε, τέθηκαν και συζητήθηκαν πολλές φορές. Φο, Υποψιάζουμε ωστόσο ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να δυναμώσουν οι γνώσεις, να ενισχυθούν οι ίδιοι ασθενείς. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα στην ενημέρωση και έχει την απέτηση στην ενημέρωση και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει να επεξετάσουμε και τι γίνεται με τις ε, δοκιμαστικές, ε, με τη διαδικασία δοκιμών. Ξέρω ότι είναι περίπλοκη η διαδικασία γραφειοκρατικά, αλλά θέλω να ρωτήσω, εξετάζει άλλες προτάσεις Επιτροπή για να ε, δει τα κριτήρια ποιότητας ε, των, της ενημέρωσης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη σαφή σας άποψη σε ό,τι αφορά τους συλλαπτήρες. Ε, υπήρχαν εδώ κάποιες ε, λα, λανθασμένες ε, απόψεις οι οποίες κυκλοφόρησαν, οπότε είναι καλό που ακούμε έτσι από ένα επίσημο πρόσωπο σαν και σας ε, αυτές τις σαφείς απόψεις. Ε, σε ό,τι αφορά την κρίση, πράγματι θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε ως ευκαιρία, ε, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της αυτοκινητομηχανίας, ο οποίος πραγματικά επλήγει περισσότερο και για τα ελαφρά λοιπόν οχήματα, όπως ανέφερε και ο κύριος Κάλαχαν, θα μπορούσαμε να έχουμε μια νέα ε, πρωτοβουλία εδώ. Αλλά ε, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν προσαρμόσει τις, ε, την φορολόγησή τους με βάση την, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ίσως λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν δεν υπάρξει πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Euro 6, δηλαδή βαρέα οχήματα, σε πρώτη ανάγνωση είχε επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά τώρα ε, προβλέπετε να αναβληθεί η σχετική ε, πρόταση. Ε, μπορείτε να πείτε κάτι. Υπήρξαν κάποιες φήμες ότι πράγματι θα υπάρξει αυτή η παράταση, ότι θα αναβληθεί δηλαδή η έγκριση της λόγω πρόταση ε, ισχύει αυτό. Και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστώ, ευχαριστήσω συγγνώμη, για τη συνεργασία που είχαμε, γιατί μπορεί να μην ήταν ε, να είμαστε πάντα τη ίδια άποψη, αλλά ήταν πραγματικά επικοδομητική συνεργασία μας και ελπίζουμε και πω ο διαδοχό σα θα ανταποκριθεί στο ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ, ήσασταν συνθετικός. Ο Κρι Ντέιβι. Ε, ερώτηση για τα αυτοκίνητα και τη μεθερμασία του κλίματος. Να εξηγήσω για τους νέους αδέλφους ότι ο κλιματισμός που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας είναι, είναι κάποιο παράγωγο, κάποια ουσία που σχέση με το υδρογόνο και είναι πολύ πιο επικίνδυνο, χίλιες τόσες φορές παραπάνω χειρότερο από το διοξίδιο. Γι' αυτό και το 2006 περάσαμε ένα, νομοθέτημα, σύμφωνα με το οποίο από το 2011 και μετά τα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούν ε, ε, μια πιο ήπια ουσία. Οπότε τώρα έχουμε αλλαγή στο τοπίο και θα πρέπει επομένω να συμμορφωθούν οι αυτοβιομήχανοι. Και όποιοι αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί θα πρέπει να αποσυρθούν. Ξεδεώσα μια ανακοίνωση επιβεβαιώντας όλα αυτά πριν από λίγους μήνες. Τώρα όμως μας λένε οι βιομηχανοί ότι αυτό το προϊόν δεν θα έχει μπει στην αγορά το 2011. Αυτό γίνεται γιατί δεν έγιναν οι αναγκαίες παραγγελίες. Δεν θέλουν να επενδύσουν οι βιομήχανοι σε αυτή την ουσία. τι, παίζουν παιχνιδάκια μαζί μας. Προβληματιζόμαστε πάρα πολύ, γιατί αυτό αφορά την υπερθέρμανση του κλίματος, επίτροπε. Ε, αυτό είναι σαν να παίζει κανείς πόκερ. Και το θέμα πιανού η μπλόφα θα περάσει. Εάν κάνει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε τα πάντα μπορεί να συμβούν. Και δεν θα πιαστώ τόπο κανένα νομοθέτημα για το κλίμα. Οπότε εσείς θα κάνετε ένα μπροστά ούτως ώστε να ξεσκεπαστεί η πλάθα τους και έτσι να χρησιμοποιηθεί αυτή η ουσία μέχρι το 2011. Κύριε Χάση, ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά το ΡΙΤΣ. Κύριε Πίτροπε, μιλήσατε για την χρηματοδότηση τη υπηρεσία για τις χημικές ουσίες. Σύμφωνο μαζί σα και εγώ ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει νομοθεσία αλλά να μην υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να εφαρμόσει η νομοθεσία η υπηρεσία. Δεν είναι ωστόσο αποδεκτό ούτε η αποδυνάμωση της νομοθεσίας κατά τη φάση της υλοποίησής της. Και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει με τον λεγόμενο κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία της νομοθεσίας ε, ρίς. Είναι οι ουσίες που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ε, καρκινογόνες, ε, τοξιογόνες ή μεταλλαξιογόνες και που σύμφωνα με την ε, νομοθεσία έπρεπε να λάβουν άδεια πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης ή υπάρχουν ήδη 800 τέτοιες ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνες ε, ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, ενώ πολλές δεκάδες ουσίες είναι γνωστές ότι δεν είναι τέτοιες. Στον κατάλογο των υποψηφίων ωστόσο υπάρχουν μόνο 15. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν εκατοντάδες ε, καρκινογόνες ισίνες, ε, ουσίες που ε, φτάνουν στο καταναλωτή. Όταν αγοράζεις, ας πούμε, ε, σεντόνια. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς αν τα σεντόνια περιλαμβάνουν ή όχι καρκινογόνες ουσίες. Αλλά το δικαίωμα αυτό δεν υλοποιείται γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής των οποίων προείσεστε εσείς κύριε Φερχόγγιν, είναι αυτές που εμποδίζουν την επέκταση του καταλόγου των υποψηφίων στις γνωστές καρκινογόνες ε, και λοιπά Γιατί. Γιατί μπλοκάρετε την επέκταση των ουσιών αυτών. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πρώτα και ευχαριστώ κύριε Πετρόπε. Ε, σε ό,τι αφορά το Eco Design ε, συμφωνώ απολύτως ε, μαζί σας ότι δηλαδή έχουν ε, ε χρησιμοποιηθεί πολύ ε, επιχειρήματα στην αλλά και στην Αυστραλία έχει γίνει μια αντίστοιχη απαγόρευση ε, γιατί ήξερε κανείς πως όποιος ε, ε, έρθει σε αντίθεση με την κυβέρνηση θα έχει να κάνει για παράδειγμα και με τον Σουατζενέγκερ εδώ πέρα. Άρα λοιπόν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι είχαν εκπροσωπηθεί και στην Επιτροπολογία είναι κάτι τέτοιο το, το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εμεί απευθύνουμε έκκληση στι κυβερνήσει να ε, πληρούν τα όσα συμφώνησαν από κοινού μαζί σα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ε, ελαφρά ε, επαγγελματικά ε, το ότι θα υποβάλει μια νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει ότι του χρόνου θα πρέπει όλοι να αγοράσουν νέα οχήματα. Πάντα προβλέπεται μια μεταβατική περίοδο, οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τα σχετικά επιχειρήματα. Τρίτον, ε, πακέτο φαρμακο, φαρμακευτικό. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ λόγω ε, του λίγου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μα σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των ασθενών. Πράγματι υπάρχουν ε, κάποιε διαφορέ ε, ε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, οπότε θα πρέπει να το γνωρίζετε κι εσεί και να το κοινοποιήσετε στον διαδοχό σα, αλλά ας α πούμε ότι δεν επιθυμεί κανεί διαφήμιση, αλλά η Επιτροπή προτείνει να αλλάξουμε τον ορισμό στο 1-3 πάντα αναφερόταν ενημέρωση και διαφήμιση ε, και εκεί υπήρξε μια διαγραφή. Αλλά το ότι αλλάξαμε απλά τον ορισμό δεν σημαίνει ή δεν αποτελεί εγγύωση ότι δεν θα υπάρχει πλέον διαφήμιση. Ανεμέρωση από την πλευρά του κατασκευαστή μέσω μέσων ε, ε, έντυπων μέσων ή άλλων μέσων ενημέρωση προφανώ και αποτελεί αυτό καθε αυτό. Μπορεί να αποτελέσει, σε πάση περιπτώσει, διαφήμιση. Άρα λοιπόν συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρίσο, οπότε ε, σχετική ενημέρωση δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο ε, μέσω τη αλυσίδα επιχείρηση φαρμακομηχανία προ καταναλωτή, αλλά ενδεχομένω να έχουμε και κάποια άλλη ουδέτερη υπηκή, ούτω ώστε να φτάσουμε ταχύτερα ε, στον στόχο που θέλουμε. Ταχύτερα από ό,τι αν δηλαδή θα έχουμε μόνο τον ένα αυτό τρόπο. Ο κύριο Πανιόλ Κύριε Αντίποδο, ευχαριστώ που κάνετε μια βολονταριστική παρέμβαση στην ομιλία σας. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική σε έναν κόσμο οικονομικής απορρίθμισης, όπου που κυριαρχούσε στο πακέτο των φαρμάκων και όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Όταν ασχολούμεθα, όπως κάποιοι συνάδελφοι είπαν νωρίτερα, στο θέμα της ε, απομίμησης φαρμάκων, έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν εφαρμόσαμε κανένα από τους νόμους που πρέπει να εφαρμόσουμε ως χωροφύλακες. Και τελικά, οι, φαρμακε... οι φαρμακοβιομηχανίες, μιλήσατε στο ξεκίνημα για την νόμιμη αλλά και την παράνομη αλυσίδα και διαπιστώνουμε κάθε φορά ότι υπάρχει ένα ξεκίνημα της Παρασκευής. Πώς Είπατε θα ξεκινήσετε επαφές με άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς. Πώς θα ξεκινήσετε αυτές τις επαφές για να ρυθμίσετε αυτή την Παρασκευή όπως έπρεπε. Παρασκευή των οποίων τα θύματα δεν είναι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες όπου εκατομμύρια ατόμων εκτός Ευρώπης. Δεύτερη, δεύτερη ερώτηση, σύντομα. Αυτές οι περιοχές σκιάς, αυτές οι ζώνες, ε, οι σκούρες ζώνες, ε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του ασθενούς. Ο ασθενής είναι μόνος. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να προστατευτεί. Είπατε κι εσείς, εισαγωγικά, ότι είναι αντικείμενο μιας μόνιμης, ε, διαφήμιση από τους ιατρικού ειδικού. Και θα έπρεπε να προστατευτεί. Ευχαριστώ. Κύριο Μπάικο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συχνά μιλούσαμε για την διαφήμιση γιατί αυτά ε, στα φάρμακα, διότι αυτό, αυτή η δραστηριότητα έχει τεράστια κέρδη. Οι παράνομες ε, δραστηριότητες στα φάρμακα οδηγούν ε, τον ασθενή να, να, να χρησιμοποιήσει φάρμακα που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Κάτι, ένα από τα χειρότερα προβλήματα του, που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη ζωή. Πιστεύω ότι τη ζωή των ασθενών πρέπει να την προσέχουμε στην Ευρώπη και πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και της διανομής των φαρμάκων. Είναι πολύ επικίνδυνη η διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης πιστεύω. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά παράδειγμα τι πω, τα φάρμακα για τη μείωση του βάρους για τη, δίαιτα, πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα πρέπει να πηγαίνουμε σε γιατρούς για να είμαστε βέβαιοι. Προφανώς υπάρχουν διαφορές, πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια μέση οδό. Δεν μπορούμε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες να καθορίζει όλους τους κανόνες για τη διαφήμιση ή την ενημέρωση σε όλη την Ευρώπη. Χρειάζονται να στηριχθούμε στην επιστημονική ε, τεχνογνωσία, αλλά θα μπορούσαμε να προτείνουμε κώδικες διοντολογίας στα μέσα ενημέρωσης που θα επιτρέπουν να τους γνωρίσουμε τις αρχές που θα είναι υπεύθυνε για την υιοθέτηση τέτοιων νόμων. Ε, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να υποστηρίξω σχεδόν σε όλα τα σημεία που έθεσε, αλλά ε, σε ό,τι αφορά την αρχή για τα χημικά, ε, ε, και για την οποία θα πρέπει να επιλύσει το σχετικό ζήτημα που έχει προκύψει, αλλά και σε σχέση με το ΡΙΤ ε, και σε σχέση με τα αυτοκίνητα και σε μια σειρά από άλλα σημεία πάντα ε, υπάρχουν αντιθέσει μετά με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, και αυτό συμβαίνει επειδή, όπω είπε ο Πέτρε επειδή συμβολούν κάποια πράγματα εδώ στο Συμβούλιο και μετά όμω όταν πηγαίνουν σπίτια τους έχουν διαφορετική στάση αυτό νομίζω θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε εάν έδινε μεγαλύτερη δημοσιότητα στις δικέ της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ το βίωσα αυτό στο Ρίτς, ε, δηλαδή μας έδωσε χίλια σελίδε ο, ο Επίτροπος και ε, επέτρεψε στου διευθυντές τους να κάνουν κάποιες παρουσιάσει, αυτό έγινε. Αλλά αυτό ε, και τίποτα παραπάνω, αλλά αυτό δεν έφτανε και βέβαια εμεί παραπονεθήκαμε γι' αυτό επανειλημμένα. Ε, και βέβαια αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει και με τη δημοσιότητα, δηλαδή και το ποια στάση θα πρέπει να λάβει ένα της ε, Ευρώπης και ούτω καθεξής ε, ως πολιτικός. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δικό μου μήνυμα, δηλαδή σε σχέση με τα όσα είπατε κύριε Φαχοήτη είναι όλα τα θετικά. Εάν οι βιομηχανίε στη δική μου χώρα και σε όλε τι υπόλοιπε χώρε, εάν δεν έχουν κεφάλαιο στη διάθεσή του, τότε θα πρέπει να κάνετε κάτι δραστικό στον χρηματοδοτικό τομέα. Και εγώ δεν ε, μιλάω ως κάποιος ξένος. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι και σας λέω δεν έχουμε τα κεφάλαια, δεν μας δίνει κανείς τα κεφάλαια. Για να μπορέσουμε τελικά να ε, προβούμε και στην ε, ανάληψη κάποιων έργων από τη δική μας πλευρά ως εταιρεία που και στον χώρο του περιοχή. Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήταν τόσο ε, ειλικρινή στο θέμα της ενημέρωσης. Και εγώ όμως έχω κάποιες επιφυλάξει όπως και άλλοι για το θέμα αυτό. έχω δουλέψει στον κλάδο αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να ενημερώνονται όσο γίνεται περισσότερο οι ασθενεί. Αυτό είναι σίγουρο. Όμω η ποιότητα τη πληροφορία επίση είναι κάτι το σημαντικό, ακριβώ όπω και το να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα ο ασθενή. Το είπατε και εσεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανεί τη διάκριση μεταξύ διαφήμιση και ενημέρωση. Ακόμη περισσότερο λόγω του εμπορικού χαρακτήρα αυτών των ενεργειών, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ε, ουδέτερη, αξιόπιστη πληροφόρηση, ε, αντικειμενική, αμερόληπτη. Και όλα αυτά τα λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν αρκεί να λέει κανένα δημοσιογραφικά ότι πρόκειται για ένα μήνυμα από την φαρμακοβιομηχανία και αυτό να θεωρείται αρκετή ενημέρωση για τον ε, ασθενή. Ε, πρέπει κάπως να ξέρει ποιο είναι το πιο κατάλληλο φάρμακο ο άλλος. Και φυσικά και η φαρμακοβιομηχανία θα πρέπει να σέβεται μια τέτοια διοντολογία. Και ξέρω τι σας λέω. Τους ε, ε, είναι λυπηρό το γεγονό ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και άλλο ε, μαζί σα ε, στο μέλλον, γιατί πραγματικά είστε ένα οραματιστή. Μπορεί να διαφέρουν οι απόψει σα μερικέ φορέ, αλλά πραγματικά έχετε οράματα. και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο έχουμε εδώ και σε κεντρικό. έχουμε εστιάσει στο ζήτημα τη δημόσια αγία. γιατί θέλουμε όχι μόνο ποσοτική ανάπτυξη, θέλουμε ποιοτική ανάπτυξη. Και αυτό το λέω και στου νέου συναδέλφου. Δεν μου αρέσει το γεγονό ότι. Ε, εδώ ξαναρχίζει πάλι η συζήτηση σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών. Εδώ και χρόνια το συζητάμε. Ε, και ο κύριο να έχει εργαστεί από αυτού του ζητήματο όλα αυτά τα χρόνια και τώρα είναι δυνατόν να λέμε ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή, να τα ε, ε, διαγράψουμε όλα. Ε, δηλαδή, τι είδου δημοκρατία είναι αυτή. Ε, αν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα όπου φλιαρούμε μόνο και δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να είμαστε ανταγωνιστικοί ε, παγκοσμίω. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα ε, που άπτεται δικαιωμάτων, όχι απλά με, με ζητήματα κέρδου. Και γι' αυτό πραγματικά εξοργίζομαι όταν ξεκινάει αυτή η φλιαρία και εκ νέου συζήτηση, όταν έχουμε συζητήσει 10 φορέ όλα αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την παραποίηση των φαρμάκων, συμφωνώ με τη συνάδελφο η οποία αναφέρθηκε στο διαδίκτυο δίκτυο και ότι ε, πραγματικά εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τι προσπάθειέ μα, γιατί και μέσω αυτού υπάρχει και μεγάλο κομμάτι της ε, προώθηση των παραποιημένων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα τώρα συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει να ε, όλες οι, όλα τα μέτρα στον τομέα τη υποδομή να προσανατολίζονται και προ τον στόχο της μείωσης των εκπομπών ούτως ώστε να επιτύχουμε και την διαφοροποίηση όλου αυτού του μοντέλου στα αυτοκίνητα. Η κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Ο έλεγχος, συμφωνώ μαζί σας ότι ο έλεγχος της απομίμησης και η ενημέρωση του πολίτη είναι βασικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, ε, μπορούμε να ελέγξουμε την ε, νόμιμη αλυσίδα, αλλά μήπως σκεφτήκατε το ενδεχόμενο να ενημερώνεται τους πολίτες, να μην αγοράζουν από το ίντερνετ φάρμακα ή τέλο πάντων να υπάρχει μια μεγαλύτερη ενημέρωση για το πώς λειτουργεί η αγορά μέσω ίντερνετ. Οι πληροφορίες, ε, οι πληροφορίες ε, που ρυθμίζονται αυτή τη στιγμή ε, από την οδηγία του 2003 προσθέτει, έχει περιλαμβάνει 24 σημεία. Ας ας εντάξουμε ένα ακόμα σημείο, ούτως ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο ασθενή να επικοινωνήσει απευθεία με τη βιομηχανία για να καλύψει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσαρμοστεί η ενημέρωση στο κάθε, ε, στα διάφορα επίπεδα του ασθενούς, στι διάφορε κατηγορίε του ασθενούς. Εγώ πιστεύω ότι η ενημέρωση πρέπει να χορηγείται από τον επαγγελματία και η γενική ενημέρωση να περιορίζεται σε ενημέρωση που θα απευθύνεται στο μέσο επίπεδο του ασθενούς. Ευχαριστώ. Η Λίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις για τα πακέτα, για το φαρμακευτικό πακέτο, το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών ιδίω. Είπε η κυρία Ρίστε ότι χρειαζόμασταν ανεξάρτητη ενημέρωση. Και αυτό είναι το ζήτημα. Ποιο πληροφορεί. Συζητούσαμε σήμερα το πρωί για τα αυτοκίνητα. Όταν θέλω να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, δεν πάω στην εταιρεία που κατασκευάζει, αλλά σε έναν ουδέτερο, ένα καταναλωτικό, ε, μια, μια οργάνωση καταναλωτών. Δεν, δεν παίρνει αξιόπιστε πληροφορίε από αυτό που σου φτιάχνει το προϊόν. Πρέπει να προσφύγει σε έναν εξάρτητο όργανο. Το πώ θα γίνει αυτό είναι δύσκολο. Αλλά αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την οδό θα υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις. Να ζητάμε δηλαδή από τις φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν ουδέτερες πληροφορίες στον ασθενή. Δεν το πολύ πιστεύω. Δεύτερο θέμα. Μιλήσατε, δεν μιλήσαμε μάλλον πολύ, για την οδηγία για την φαρμακοεπαγρύπνηση σήμερα. Είμαι εισηγήτρια. Αυτό που βασικά ήθελα να πω είναι ότι αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Ενώ στο Συμβούλιο το θέμα που συζητείται είναι ποιο θα είναι σε κάθε επιτροπή. Αν θα είναι ένα από κάθε κράτο μέρο τη επιτροπή ειδικών. Αλλά η έμφαση θα πρέπει να είναι λειτουργεί το σύστημα. Καθίστανται ασφαλή τα φάρμακα για τον ασθενή. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπατε προηγουμένω, κύριε Επίτροπε, για την οδηγία REACH. Ε, δεν, είναι, δεν έχει νόημα να ζητούν οι κυβερνήσει, να υπάρξει ένα πολύ ε, σύνθετο σύστημα στην Ευρώπη και να μην χορηγούν κατόπιν στο σύστημα αυτό τα κονδύλια για να λειτουργήσει σωστά. Η βάση δεδομένων τώρα για την φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να έχει κονδύλια, προσωπικό και έμφαση. Και άρα θα πρέπει και θα πρέπει να ξαναγυρίσει σαν, να έχει σαν βάση της, σαν κέντρο της, σαν έμφασή της τον ασθενή. Λυπούμε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει. Μη θυμώσετε. Μαζί μου. Θα σας δώσω προτεραιότητα στην επόμενη συνάντηση. Κύριε Φερχόγγεν, πολλές ερωτήσεις. Τι απαντήσεις έχετε και αν μπορούν οι διερμηνείς να μας δώσουν και πέντε λεφτά ακόμα. ξέρω. το γεγονό ότι τόσοι πολλοί ε, συνάδελφοι θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Να πω καταρχήν ότι πράγματι ναι, υπάρχουν προβλήματα με του. Ε, με τα κράτη-μέλη και με λύπη μου διαπιστώνω ε, το γεγονός αυτό και θεωρώ μάλιστα πως ε, δεν θα επιτύχουμε και κάποια περαιτέρω πρόοδο στο πλαίσιο της ειδική ε, προεδρίας καθώς δεν έκανε κάποια περαιτέρω κίνηση, δεν έλαβε χώρα ούτε μία ε, συνεδρίαση υπό τη Σουηδική Προεδρία για αυτό το ζήτημα και θα έχω τη δυνατότητα να συζητήσω αυτό το ζήτημα μαζί της. Ε, πίσω από αυτήν την ε, προσέγγιση της κρύβεται ένα, μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων μεταξύ των κρατομελών σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών. Και εδώ υπενθυμίζω για συνταγογραφούμενα φάρμακα, για να μην συχαίουμε λίγο τα όσα συζητάμε. Μιλάμε πάντα για συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ε, σε κάποια λοιπόν κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις γιατί θεωρούν πως ε, ένας πιο ενημερωμένος ασθενής τι συνεπάγεται υψηλότερο κόστος. Ε, αλλά εγώ δεν θεωρώ πως υποχρεωτικά κάτι τέτοιο θα λάβει η χώρα. Εμείς έχουμε μία μελέτη από την αρμόδια αρχή μας στο Λονδίνο, η οποία μελέτη εκπονήθηκε με βάση την παραμονή στο νοσοκομείο ασθενών οι οποίοι είχαν ε, νοσηλευθεί λόγω της λήψης λανθασμένων φαρμάκων και ε, να μην εκπλαγείτε αν σας πω ότι το 5% των ασθενών που βρίσκονται στα βρετανικά ε, νοσοκομεία ε, βρίσκεται εκεί γιατί ακριβώς είχε ε, λάβει ένα λαθασμένο σκεύασμα, δηλαδή αν ήξερε τι να λάβει αυτό το 5% δεν θα βρισκόταν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και από προληπτικής άποψης και κατά συνέπεια και από άποψης μείωσης του κόστους. Άρα λοιπόν η γραφειοκρατία των κάποιων κρατών μελών, ειδικότερα ε, της χώρας στην οποία εγώ γνωρίζω καλύτερα, ε, έχει αντιταχθεί, πράγμα το οποίο βρίσκω πολύ περίεργο. Άρα λοιπόν, ε, εκείνο που ε, πρέπει να πω είναι πως ο αγώνας ε, κατά της γραφειοκρατίας των Βρυξελών είναι δύσκολος αλλά είναι δυνατόν να κερδιθεί ενώ ο αγώνας κατά της γραφειοκρατίας των κρατών μελών στον χώρο της υγείας είναι δύσκολο να κερδιθεί, σχεδόν αδύνατο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα, σε ό,τι αφορά το Euro 5 και Euro 6 θα επιμείνουμε, θα παραμείνουμε στα όσα έχει σκοπό να προβλέψει ο νομοθέτηση. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή κάποια πρόταση νομοθετική ε, ή οτιδήποτε άλλο, κάποια παράταση. Όχι, οι κατασκευαστές θα πρέπει να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν ξέρω από πού ε, προέρχεται αυτή η συζήτηση την οποία έθιξε ο κύριος Παλαισκής. Δηλαδή, ε, κάποιοι κατασκευαστές λένε ότι δεν είναι διαθέσιμα τα οσα εχουν συμφωνηθει δεν ξερω απο που προερχεται αυτη η συζητηση την οποια εθιξε ο κυριος παλαιστης δηλαδη καποιοι κατασκευαστες λενε οτι δεν ειναι διαθεσιμα τα αντιστοιχα ε, ανταλλακτικά ε, και γνωρίζουμε ότι πράγματι δεν, έχουν, ε, δεν τα έχουν παραγγείλει γιατί δεν ήθελα να ξεκινήσω τη μαζική παραγωγή. Να σας πω, το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Εάν κάποιος δεν τηρήσει τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις, τότε ισχύουν τα όσα έχουμε προβλέψει τότε, για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος ε, θα, ε, σε ένα κράτος μέλος ο καταναλωτής ε, θα κληθεί είτε να αγοράσει ένα παλαιότερο αυτοκίνητο είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς κλιματιστικό μέσα. θα δούμε το πώς έχει η κατάσταση μέσα στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό αφορά μόνο τη δική μου περιέργεια, γιατί πραγματικά είμαι πεπισμένος ε, πως ε, θα υπήρχαν οι αντίστοιχες επενδύσεις από την πλευρά των κατασκευαστών εάν υπήρχαν και αντίστοιχες παραγγελίες. Εν πάση περιπτώσει είναι υποχρεωμένοι ε, οι κατασκευαστές να τηρήσουν τα όσα έχουν προβλεφθεί. Κυρία Χάση, τώρα να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα ή κάποιο κάποια προσπάθεια να μην ισχύσει με τον τρόπο που πρέπει και να ενημερώνονται με τον τρόπο που πρέπει ο κατάλογος των υποψηφίων. Ε, ε, σεβασμάτων, ε, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι θέλουμε πραγματικά να μας προστατεύσουμε από καρτινογόνες ουσίες οι οποίες επηρεάζουν και την αναπαραγωγική ικανότητα αλλά και τις μεταλλαξιογόνες ουσίες. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εδώ να έχουμε δεσμεύσεις. Έχουμε τακτικότατη ενημέρωση και συμπερίληψη στο κατάλογο των υποψηφίων ουσίες και έχουμε και μία σειρά από ουσίες για τις οποίες ήδη έχουμε προβλέψει επαγόρευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κύριο Βίζε, ε, πράγματι θα συμφωνήσω με τα όσα ανέφερε ως προστάση των πολιτικών στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ. Και σε ό,τι αφορά τις ε, αξιώσεις απέναντι στη βιομηχανία, θα πρέπει αυτές να τις θέσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Και δεν είπα ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πρόταση, απλά σα είπα πω οι προθεσμίε τι οποίε θα προβλέψουμε μέσα σε τέτοιες προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη του και τι επενδυτικέ δυνατότητε από την πλευρά ε, τη βιομηχανία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δεν έχει καθόλου δυνατότητα να προβεί σε νέες επενδύσεις η αυτοκινητοβιομηχανία. Θα το σκεφτούμε λοιπόν αυτό το ζήτημα όταν τα φτάσουμε και άλλα, δεν απέχει πολύ αυτό το σημείο. Κύριε Λίζε, ε, δεν είναι σωστό αυτό που είπατε ότι δηλαδή άλλαξε απλά κάτι στον ορισμό ε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών. Προφανώ έπρεπε να αλλάξει ο ορισμό όταν λέγαμε και ενημέρωση και διαφήμιση. Γιατί θέλουμε να επιτρέψουμε ενημέρωση χωρί να θέλουμε να επιτρέψουμε διαφήμιση. Ε, διαπίστωσα σε ένα μέσο ενημέρωση γερμανικό, ε, για κανάλι μιλάω τηλεοπτικό, να αναφέρεται πώ η Επιτροπή επιθυμεί διαφήμιση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων και αυτό το βασίζει απλά σε ένα κείμενο το οποίο λέει η ενημέρωση ε, η διαφήμιση σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους συσκευάσματα απαγορεύεται. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν τι ακριβώς ε, σκέφτονται, πώς φτάνουν σε τέτοια συμπεράσματα τόσο αυθαίρετα. Εγώ λοιπόν έχω σπουδάσει δημοσιογράφος και δεν θα θεωρούσα πως υπάρχει καθόλου δημοσιογραφική ηθική σε αυτόν τον κόσμο, εάν μου έλεγε κανεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει σαφή διαχωριστική, διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωση αφενό και διαφήμιση αφετέρου. Αυτό το κάνουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι στη δουλειά του και είναι ήδη σαφέ το τι συνιστά τελικά διαφήμιση και τι δεν συνιστά διαφήμιση. Πρόκειται λοιπόν για ένα εμβόλυμο, για ένα έολο επιχείρημα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να ε, έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ ενημέρωση και διαφήμιση. Είναι πάρα πολύ συστατική, πάρα πολύ ε, ε, μινιμαλιστική, αν θέλετε, η πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτές τις υποχρεώσεις εδώ. Μιλάμε απλά για μία έγκριση εδώ η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Και ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση, εφόσον το επιθυμεί, σε πληροφορίες οι οποίες έχουν διατεθεί ε, μετά από έγκριση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ε, μία αντικειμενική πληροφορία που έχει, που έχει χαρακτηριστεί ως αντικειμενική από την αρμόδια ελεγκτική αρχή να εκλαμβάνεται ως διαφήμιση. Ε, πάντως αυτό είμαι πολύ σαφής και δεν θα προβώ σε περαιτέρω διαβούλευση αυτό το ζήτημα. Εάν θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν να ε, ξεφύγουν από αυτό το πρόβλημα, χωρίς να προβλέψουν δηλαδή ε, συγκεκριμένες διατάξεις εδώ, ως προς τα, στα όσα είναι απαραίτητα ε, σε σχέση με την Ένωση για τα φάρμακα, τότε η ανάγκη για ενημέρωση θα αναζητήσει άλλα κανάλια πληροφόρησης και εκεί πραγματικά θα χάσουμε απολύτως τον έλεγχο. Άρα λοιπόν προσπαθούμε εδώ να μειώσουμε τέτοιου είδους αναλυτικές ε, πηγές ενημέρωσης. Κύριε Μανιώ, δεν υπάρχει τέτοιου είδους ε, ρύθμιση στον τομέα των φαρμάκων συγγνώμη, απορρίθμιση. Ε, μέχρι στιγμής ε, όλο και περισσότερο κατά τελευταία χρόνια αυστηρότερες διατάξεις έχουμε. Εάν έχετε ένα ε, παράδειγμα για προϊόντα απορρίθμιση σε αυτό το τομέα, παρακαλώ να μου το αναφέρετε. Αλλά θέσατε ένα ε, πολύ σοβαρό ερώτημα, δηλαδή του πού παράγονται τα εν λόγω φάρμακα και εδώ συνεργαζόμαστε στενά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και με άλλα του ώστε να μπορέσουμε να ε, προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε την παράνομη ε, παρασκευή φαρμάκων. Πάντως ε, σας λέω πως το φαινόμενο αυτό εντός της Ευρώπης είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή πολύ λίγες ήταν οι περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκαν πραγματικά παράνομα εργαστέρα παρασκευής. Αναφέρομαι στην εσωτερική ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστε λοιπόν περιπτώσει όπου πραγματικά ε, είχαμε τέτοια παρασκευή σκευασμάτων τα οποία προορίζονταν για την ίδια την ευρωπαϊκή αγορά. Άρα λοιπόν για το άλλο το κομμάτι, δηλαδή των σεβασμό που πραγματικά ε, βάζω το παράδειγμα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχουμε διεθνή συνεργασία. Ε, Επίση, να απαντήσω σε αυτό που είπατε, ε, δεν έχουμε να κάνουμε εμεί συνταγογραφούμενα φάρμακα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση για προϊόντα, εδώ αυτή γίνεται ούτως ώστε να πιστεί ο καταναλωτής ε, για να αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει στον χώρο του συνταγογραφόμενου φαρμάκου, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει αυτό το φάρμακο ο καταναλωτή ούτως ή άλλως. Μπορεί να το λάβει μόνο εφόσον ένας ιατρός με δική του ευθύνη συνταγογραφήσει το νόμο φάρμακο. Και σε σχέση με αυτή τη διαδικασία της συνταγογράφησης δεν αλλάξει και τίποτα. Δηλαδή η ίδια η αγοραστική αν θέλετε δύναμη τελικά και η απόφαση αγοράς δεν επηρεάζεται από την πλευρά του ασθενού, καθώ την εν λόγω απόφαση δεν την λαμβάνει όπως σας λέω ο ασθενή. κύριε ε, Φλόρεντ, ε, και ζητώ συγγνώμη που έχω αλλάξει εδώ τη σειρά των ερωτήσεων σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση της ε, βιομηχανίας σε επενδύσεις, δηλαδή τη δυνατότητά της να προβεί σε επενδύσεις ε, και τις σχετικές υποχρεώσεις που υποβάλλουμε εμείς ως νομοθέτης. Αντίστοιχα προβλήματα είχαμε αντιμετωπίσει μέσα στα στα προηγούμενα χρόνια ε, με σχετικές βιομηχανίες όπου δεν υπήρχε δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις. Για παράδειγμα θα θυμόσαστε ίσως ε, τον περσινό Οκτώβριο που είχα αναφερθεί εδώ στο γεγονός ότι θα χρειαστούμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση. Καθώς ε, ε, θεωρούσε, ήταν όλοι αρνητικοί και ήθελαν να, να πούν πως όχι δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε την αυτοκινητομηχανία. Αλλά εμείς δεν θέλαμε κάτι τέτοιο. Εμείς βλέπαμε ότι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ε, και είπαμε ότι αν θέλουμε να τηρηθούν οι διατάξεις που έχουμε προβλέψει τότε θα πρέπει να γίνουν και αντίστοιχε επενδύσει. Και με χαρά μα βλέπουμε πω ε, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεω έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο, αλλά μιλάμε για δανειοδότηση εδώ. Δεν μιλάμε για ενισχύσει, για διονότηση δηλαδή δάνεια τα οποία θα κληθούν να αποπληρώσουν οι βιομηχανίε. Με τον κύριο Χατζημαρκάτη να πω ότι συμφωνώ απολύτω. Και νομίζω πως απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τοβαχόγη. Ε, ε, σα ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σα σήμερα εδώ στην συνεδρία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Όπω είπε ο κ. Χατζημαρκάκη, είστε ένα ρομαντιστή. Ε, έτσι κι αλλιώ δεν ξέρουμε αν θα είναι η τελευταία μα συνεδρίαση η σημερινή, γιατί είπατε θα εργάζεστε μέχρι τελευταία μέρα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά. Γεια σα. Διακόπτουμε μέχρι τι 3.